Uh, ladies and gentlemen, could um, to, uh, to find... μπορούμε να καθίσουμε παρακαλώ. Έχουμε επιφανείς ομιλητές κοντά μας που άλλο δεν περιμένουν παρά να έχουν την ευκαιρία να σας μιλήσουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα έχουμε πιστεύω θέσεις αρκετές για όλους. πολλούς γνωστούς και ενδιαφέροντες βλέπω εδώ γύρω. Έχουμε την Υπουργό κυρία Νόρικα, είναι. Χρειάστηκα βοήθεια για να φέρω σωστά το όνομά σας. Ε, λοιπόν εκεί Προεδρία εκπροσωπεί. Το Μισελ Μπαρνιέ φυσικά. Ο οποίο τακτικά έρχεται στι συνεδριάσει μα. Τον καλωσορίζουμε. Θα εξηγήσω τα διαδικαστικά σε λίγο, τα οργανωτικά. Uh, so um, let's um, uh, uh, Θα κάνω μερικές ε, εισαγωγικές παρατηρήσεις. Ενώ εσείς βλέπετε την αφίσα της συνεδρίασης. Καλωσορίζω φυσικά και όλους τους ε, ε, θεατές μας από το διαδίκτυο Μην ξεχνάμε ότι ο μήνας που είναι ο μήνας της ε, ενιαίας αγοράς. Είχαμε και τηλεσυζήτηση την Τετάρτη και επέμεινα ιδιαίτερα σε αυτό. Και εδώ βλέπουμε όλη την προσπάθεια της Επιτροπής μας ώστε να οργανώσουμε περισσότερο και πιο ουσιαστικά τη δουλειά μας και στο λιανικό εμπόριο για την εσωτερική αγορά, που ασφαλώς έχει να κάνει και με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά και με την προστασία του καταναλωτή, ώστε να έχει αυτός το προϊόν που θέλει, γνώσεις για το προϊόν που σκοπεύει να αγοράσει, προστασία των δικαιωμάτων του, όλα αυτά τα θέματα που έχουν κρίσιμη σημασία, όσο κρίσιμη βέβαια έχει και η οργάνωση της αγοράς. Η προστασία, η ασφάλεια των προϊόντων, και όλα αυτά τα οποία έχουν τόσο μεγάλη σημασία για την λιανική αγορά. Όπως βλέπετε, ο τίτλος μας είναι για μια πιο αποτελεσματική και δίκαιη, ισότιμη λιανική αγορά στην Ευρώπη. Ευχαριστώ την κυρία Κοράτσα Μπίλτ που είναι εδώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ντε Ιόγκ που έχει και την έκθεση. Τη Χάντι Ρούλε, Σκιώδη και άλλους συναδέλφους που φαντάζομαι θα έρθουν αργότερα. Στόχος μας λοιπόν με την ακρόαση αυτή ήταν να επιτρέψουμε να συναντηθούν διάφοροι παράγοντες. Στόχος μας είναι η άρση των εμποδίων. Αυτό θα μας πάει μέχρι τις 4. Και μετά η ευθύνη και η ισότιμη μεταχείριση με βάση και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Μπέρι, κυρία Μπέρι, είναι εδώ παρούσες, θα μας δώσουν τις προτάσεις τους. Η Επιτροπή μας, σε μια ρηξικέλευτη προσπάθεια επικοινωνίας με τον πολίτη, έχει θεσπίσει και ένα feed Twitter με ένα hashtag που έχει τον τίτλο Retail Roundtable. Εάν λοιπόν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή μας κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως, μπορείτε να μας στείλετε τις παρατηρήσεις σας στο hashtag δίεση Retail Roundtable. και θα απαντήσουμε ζωντανά στις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Θα παρακαλέσω βεβαίως πέραν των ομιλητών, εφόσον υπάρχει χρονικό περιθώριο, και άλλους ε, ομιλητές να μιλήσουν. Εάν ε, δεν έχουμε χρόνο φυσικά θα σας περιορίσω, αλλά οποιοδήποτε θέλει να παρέμβει στη συζήτηση είναι ευπρόσδεκτος να σηκώσει το χέρι και να μου ζητήσει το λόγο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις πρώτες και εισαγωγικέ τοποθετήσεις. Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ. Θέλεις και ρολόι για να βλέπεις το χρόνο σου, έχεις πέντε λεπτά. Η Υπουργός νομίζω θα μιλήσει στο τέλος. Μετά θα ακούσουμε τον Μισελ Μπαρνιέ, θα ακούσουμε τον Ντένις Ντε Ιόγκ. Και θα παρουσιάσω και τους ειδικούς μας με τη σειρά τον καθένα. Μαρία, έχεις το λόγο με ευχαριστώ και ευχαριστώ ιδιαίτερω για την ε, απίστευτη υποστήριξη όλο αυτό το διάστημα, σε όλα αυτά τα χρόνια στη δουλειά μα. Ευχαριστώ τον Επίτροπο, χαιρετίζω την κυρία Υπουργό, του συναδέλφου, όλου ε, του ομιλητέ που είναι εδώ παρόντε και όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να ε, τοποθετήσουν στην αγορά την πολιτική αγορά της Ευρώπης το λιανεμπόριο. Προσπαθούμε λοιπόν, όπως είπε και ο Μάλκο μας, με το Συμβούλιο, το, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να διατηρήσουμε στην επικαιρότητα την πολιτική το λιανικό εμπόριο όσο χρειάζεται, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε με κάθε σοβαρότητα και προσοχή. Και εδώ μπορείτε να, να, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι βρίσκεται χώρο συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων. Τι σας απασχολεί, τι έχετε επιτύχει, τι θέλετε να επιτευχθεί. Και να δεσμευτούμε, να εργαστούμε για την ελευθερία, για μια νομοθεσία της ενιαίας αγοράς που θα ισχύει ε, σε όλη την Ευρώπη, χωρίς εμπόδια, χωρίς προσκόμματα, χωρίς περιορισμούς έτσι ώστε να μπορείτε να ε, αγγίξετε 500 εκατομμύρια πολίτες και ε, αυτά τα 500 εκατομμύρια πολίτες να μπορούν να ε, ζητήσουν τις προτάσεις σας. Έτσι λοιπόν, με ευθύνη και με έντιμο, ισότιμο τρόπο και ισότιμη αντιμετώπιση θέλουμε να λειτουργεί αυτή η εσωτερική αγορά, η εσωτερική αγορά των λιανικών, της λιανικής ε, πώλησης. Έτσι λοιπόν, χαιρετίζουμε την υπογραφή από 450 ε, διευθυντές διοικητικών συμβουλίων και προέδρων ε, διοικητικών συμβουλίων από διαφορετικές επιχειρήσεις της ε, πλατφόρμας για τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων B2B business to business. Βλέπω ότι έχετε εκπροσώπους εδώ που ενδεχομένως να αισθάνονται κάποιες ανησυχίες και ήθελα να συζητήσουν. Εγώ συμφέρει όλους να συζητήσετε, να τοποθετηθείτε, να εκφράσετε τις ανησυχίες σας, να συμμετάσχετε στην προσπάθεια αυτή ώστε να λύσουμε μαζί τα προβλήματα. Και ήθελα εδώ να σταματήσω, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε χρόνο για να ακούσουμε τους ομιλητές. Γι' αυτό παρακαλώ Πρόεδρε δώστε αρκετό χρόνο για τη συζήτηση. Ελπίζω να γίνει μια πραγματικά ειλικρινή συζήτηση. Ευχαριστώ. Βλέπετε που εμφανίζεστε και στο Twitter μας. Και οποιοδήποτε μας ακολουθεί στο Twitter μπορεί να συνδεθεί και να μας ακούσει live. Και τώρα θα κάνει την παρουσίασή του ο Μισελ Μπαγνιέ. Ήταν μια κοινή διοργάνωση της Επιτροπής μας και της Κομισιόν και ελπίζω να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Ευχαριστώ, Μάλκομ. Καλημέρα σε όλους. Με μεγάλη χαρά σας βρίσκω σε αυτό το φόρουμ που είναι δικό σας φόρουμ όπου θα εκφράσετε τις προτάσεις, ιδέες, τις επικρίσεις σας μετά από την πρόσκληση του Malcolm Harbour και της uh, κυρίας Κοράτσα Μπίλτ. Χαίρομαι για το ζήλο του, για αυτό το θέμα, που είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μείνει πάνω-πάνω στην ατζέντα. Είναι δύσκολο θέμα, θέλω να πω δύο λόγια γι' αυτό, γι αυτό και είναι και ένα σημαντικό θέμα. Είναι και υπουργό εδώ, η οποία είναι πολύ δραστήριοι για το θέμα της εσωτερικής αγοράς. Χαιρετίζω την αποτελεσματικότητα της Λιθανικής Προεδρίας ως προς το φάκελο αυτό. Ε, χαιρετίζω τους ευρωβουλευτές, τον κ. Ντεγιάνγκ, που θα πάρει και το λόγο σε λίγο. Βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή, το είπε και ο Πρόεδρος, σε ό,τι αφορά την ενιαία αγορά. Από τη Δευτέρα ξεκινήσαμε τέσσερις εβδομάδες δημόσιας συζήτησης στο ίντερνετ. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει με διαδραστικό τρόπο να ακούσει ιδέες, προτάσεις, κριτικές για τα μεγάλα θέματα της εσωτερικής αγοράς. Από κάτω προς τα πάνω. Από όλες τις χώρες και τις περιοχές της Ευρώπης. Έχουμε 24 πλατφόρμες, 24 γλώσσες. Πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο. Ούτω ώστε να μην μπλοκάρουμε κανένα λόγω του προσκόμματο τη γλώσσα. Και, όλες τις... και κάθε εβδομάδα για, την... για τα κοινωνικά θέματα, για την απασχόληση, για την ψηφιακή αγορά. Θέλω να πω δύο λόγια. Και για τη σχέση των πολιτών με τις τραπεζές τους. Αυτά ήταν τέσσερα μεγάλα θέματα. Ξεκινάω τη συζήτηση και χαίρομαι πάρα πολύ. Ξεκινάει μάλλον η συζήτηση και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το μήνα διαλόγου θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Εδώ δεν έρχομαι για να σε εξηγήσω ότι όλα τα ωραία και υπέροχα και θαυμάσια πράγματα που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει ό,τι κάνει μόνη της. Υποβάλλει κείμενα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Και εκείνοι βελτιώνουν τα, μας, τα κείμενά μας τα κείμενά μας πρέπει να επικριθούν, πρέπει να υπάρξει αντιπαράθεση, πρέπει να ακούσουμε ιδέες. Το λέω αυτό και στο Συμβούλιο. Και είναι σημαντικό σήμερα να ξεκινήσει η συζήτηση. Πέρα από το μήνα για την ενία αγορά, πρέπει να πούμε ότι δεν βγήκαμε από την οικονομική κρίση, δεν βγήκαμε από αυτό το τούνελ ακόμα ή από την κρίση εν γέννη. Παρότι κάναμε πολλά σωστά πράγματα για να ξαναβάλουμε την Ευρώπη στη σωστή τροχιά, σε παράλληλη τροχιά, σε παράλληλε τροχέ, όπω ακριβώ αυτέ τι δύο που, πάνω στι οποίε κινούνται τα τρένα. Η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης βελτιώθηκε, η κάθε χώρα δουλεύει για να διαχειρίζεται καλύτερα τα δημόσια οικονομικά της. Οι βάσεις της οικονομίας μας γενικά είναι πιο σταθερές. Το τρένο ξαναφεύγει από το σταθμό. Είναι η πρώτη μάχη αυτή. Και για να συνεχίσουμε πρέπει να δώσουμε τη μάχη της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Σε αυτή τη μάχη, εγώ νομίζω ότι κάθε πολίτης είναι απαραίτητος, κάθε επιχείρηση είναι απαραίτητη, κάθε περιοχή της Ευρώπης είναι απαραίτητη. Έχω αυτή την πεποίθηση, το λέω. Τώρα, το θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει σήμερα, αυτό το, αυτός ο οικονομικός τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκπροσωπεί 6 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μερικές φορές είναι και μεγαλύτερες και πάνω από 18 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Κάθε πολίτης, κάθε επιχείρηση, κάθε περιοχή συνεισφέρουν. Ε, αυτός το ήταν από τους κινητήριους της ανάπτυξής μας, πρέπει να παραμείνει και να βελτιώσουμε τη θέση μας. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε τις νέες προκλήσεις που οι επιχειρήσεις αυτού του παραδοσιακού, όπως λέμε, τομέα προσκρούν κυρίως το, την πρόκληση που αντιμετωπίζει ο έμπορος. Πρέπει, θα, θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτόν τον τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές και νομίζω ότι η λιανέμπορη δεν είναι απλώς μια ενδιάμεση, ένα ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στον προμηθευτή και στον καταναλωτή. Γι' αυτό ακριβώ η Κομισιόν τον Ιανουάριο ξεκίνησε το σχέδιο δράση για το λιανεμπόριο, βασιζόμενοι στι συστάσει και στι ιδέε τη Άννα ε, Μαρία Κορατσαμπίλτ, προ, προτείνοντα κάποια πράγματα για την ανταγωνιστικότητα του τομέα, για να καταπολεμήσουμε κάποια εμπόδια και δυσκολίε επίση. Προωθήσαμε την εφαρμογή αυτού του σχεδίου και ακριβώ γι' αυτό δημιουργήσαμε μια ομάδα υψηλού επίπεδου για το λιανεμπόριο για να εμβαθύνει σε αυτή τη στρατηγική και να την προσαρμόσει σίγουρα. Θα αρχίσει να συνεδριάζει πολύ σύντομα, δηλαδή η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει το Δεκέμβριο, για να δώσει ιδέε στην Κομισιόν, για να έτσι, φέρει μια κριτική ματιά στις δικές μας προτάσεις και προσανατολισμούς. Τώρα, η στρογγυλή τράπεζα που ξεκινάμε σήμερα, αυτή η ομάδα υψηλού επίπεδου για την ανταγωνιστικότητα του λιανεμπορίου που θα ξεκινήσει να, δημιουργεί, να συνεδριάζει, καθώς και το φόρουμ ψηλού επίπεδου για την αλυσίδα νεφοδιασμού, Δεν δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα, αυτά τα φόρουμ, αυτά τα βήματα για τα θεσμικά όργανα, για μας. Εμείς είμαστε στην υπηρεσία σας για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Αυτές οι ομάδες, αυτές, αυτά τα φόρουμ δημιουργήθηκαν για τους καταναλωτές, για τους λιανεμπόρους και για τους προμηθευτές, ούτως ώστε το σύστημα αυτό να λειτουργεί πιο εύρυθμα και να φύγουν, να εκλείψουν κάποιες δυσκολίες. Εξού λοιπόν και η δουλειά που θα κάνουν αυτά τα διάφορα βήματα, αυτά τα φόρουμ, θα είναι συμπληρωματική. Και σκοπός είναι να βελτιωθεί η θέση όλων των παραγόνων στην αλυσίδα αυτή. Μην ξεχνάμε και τη δουλειά μας του κύριου Ντεγιούγκα, ο οποίος είναι εδώ, τον οποίο ευχαριστώ, ο οποίος συνεισέφερε πολύ για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το τομέα και τις δράσεις που πρέπει να προωθήσουμε για τα ευαίσθητα θέματα. Τώρα σας σκιαγράφησα καταρχάς το πλαίσιο. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας δύο λόγια για τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Καταρχάς, το θέμα των αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Είναι το πιο λεπτό και ευαίσθητο θέμα, το δίχως άλλο. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που κάναμε στα πλαίσια της Πράσινης Βίβλου μας έδωσαν, μας φώτισαν, μας διαφώτισαν για αυτό το πρόβλημα και προέκυψε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν αυτές οι πρακτικές, ότι είναι πολύ σοβαρές. Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις, διάφορες πολεμικές θα έλεγα, για τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται αυτές οι πρακτικές, για τις επιπτώσεις τους. Και γίνεται διαφορετική ανάλυση από τους ΜΕΝ και τους ΔΕ για τον τρόπο που μπορούμε να μειώσουμε αυτές τις πρακτικές και για να τις καταπολεμήσουμε. Ε, πολλοί προμηθευτές και σχεδόν όλοι οι λιανέμποροι αναγνώρισαν την χρησιμότητα της εθελοντικής ε, πρωτοβουλίας ε, που βασίζεται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών. Πολλοί προμηθευτές, ειδικά οι γεωργοί, οι παραγωγοί, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζητούν αυτή την συμπληρωματική, αυτή την ε, πρωτοβουλία να τη συμπληρώσουμε με μια ανεξάρτητη αρχή, όπως υπάρχουν σε πολλές χώρες. Υπάρχουν αυτές λοιπόν οι ανεξάρτητες αρχές που εποπτεύουν τόσο ώστε να εφαρμόζονται σωστά οι κανόνες. Έχουν ερευνητικές αρμοδιότητες. Εμένα με ενδιαφέρει η αξιολόγηση που κάνουν αυτές οι αρμόδιες οι ε, ανεξάρτητες αρχές, αρχές στις χώρες όπου υπάρχουν. Πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα που θα μπορούσαμε να τη γενικεύσουμε. Αυτή η εθελοντική πρωτοβουλία οπωσδήποτε μπορεί να παίξει ένα ρόλο από την πλευρά της. Ε, διαπιστώσαμε ότι πολλές επιχειρήσεις ε, πήραν μέρος σε αυτήν την πρωτοβουλία, ε, επένδυσαν σημαντικούς πόρους ούτως ώστε να λειτουργήσει καλά και αυτό είναι καλά μαντάτα. Υπάρχουν όμως και άλλες προκλήσεις. Όσοι συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία θα πρέπει να αποτελούν μια μεγάλη έτσι, πλειάδα, να, να αποτελούν μια κρίσιμη μάζα από όλα τα κρατη και να εκπροσωπούν όλη την αλυσίδα ανεφοδιασμού. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια καλή εκπροσώπηση. Αυτό δεν το έχουμε πετύχει. Την αντιπροσωπευτικότητα αυτή δεν την έχουμε πετύχει ακόμα, παρότι υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί ας πούμε, φορείς και τα λοιπά από τον τομέα της παραγωγής, της μεταποίησης ή της κατανάλωσης. Θέλουμε όμως μια αντιπροσωπευτικότητα σε όλα τα επίπεδα. Οι γεωργοί που είναι η της καταναλωσης θελουμε ομως μια αντιπροσωπευτικοτητα σε ολα τα επιπεδα οι γεωργη που ειναι η βαση και που με την εργασία τους δίνουν πολλά στοιχεία ε, δεν είναι απόλυτα πεπισμένοι για αυτή την πρωτοβουλία. Δεν τους έχουμε πείσει 100%. Θέλω να δημιουργήσουμε ένα πνεύμα έτσι, συνεργασίας, εμπιστοσύνης, γιατί δεν θα ήταν αξιόπιστη αυτή η πρωτοβουλία εάν ο γεωργικός τομέας δεν συμμετείχε, αν δεν έβρισκε τη θέση του σε αυτή την πρωτοβουλία. Επίσης, για να είναι αποτελεσματική αυτή η πρωτοβουλία, θα πρέπει να γίνει και πραγματικότητα σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό η συμπληρωματικότητα με τις εθνικές ε, εθελοντικές πρωτοβουλίες και η δημιουργία ε, εθνικών, ε, εθνικής πλατφόρμας όταν δεν υπάρχει είναι απαραίτητα στοιχεία για να συμπληρώσουμε το πλαίσιο αυτό και τις προσπάθειες που κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προσπάθειες να καταπολεμήσουμε τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές δεν θα τελειώσουν με την υλοποίηση αυτής της εθελοντικής πρωτοβουλίας η δράση που πρέπει να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε με αμήλικτο τρόπο αυτές τις πρακτικές είναι σημαντικές, αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Νομίζω ότι οι υπεύθυνοι, τα κράτη-μέλη, οι κομισιόν, υπεύθυνοι της πρωτοβουλίας, θέλω να πω, οι κομισιόν, τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν πολλά πράγματα κόμμα πρέπει να ενισχύσουν αυτή την πρωτοβουλία για να εξασφαλίσουν το σεβασμό των κανόνων χάρη στην αρμόδια αρχή που υπάρχει σε ορισμένες χώρες και που έχει τις κατάλληλες αρμοδιότητες, εποπτικές αρμοδιότητες. Το θέμα δεν είναι αν η καλή οδός είναι η νομοθεσία ή η αυτορύθμιση. Από τη δική μου θέση, από το δικό μου φόκο, το μόνο που, θέλ, που θέλω και εύχομαι είναι να λειτουργήσει το πράγμα. Λέω συχνά στην Αναμαρία ότι το συμβόλιο είναι καλύτερο από την επιβολή. Ο θελοντισμός, δηλαδή, αν η σύμβαση είναι πιστική, αν πούμε δηλαδή ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι στηρίζεται από πολλούς φορείς και τα λοιπά, υπάρχει την προσωπευτικότητα και πείθει τον κόσμο και τότε και εγώ από πλευράς Κομισιόν θα βγάλω ε, κάποια συμπεράσματα. Ελπίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία θα λειτουργήσει. Εμείς από την πλευρά μας, από την πλευρά μας θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Επίσης κάνουμε και μια ανάλυση, μια μελέτη αντικτύπου. Και θα πάρουμε και μια απόφαση φέτος για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά οι προσπάθειές μας δεν τελειώνουν εδώ. Αυτά ήθελα να σας πω για μένα, για τους συναδέλφους μου. Στο τέλος αυτών των αρχικών παρατηρήσεων θα πρέπει να φύγω δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, ο ένας επικεφαλής, ένας ε, εκπρόσωπος από το γραφείο μου είναι εδώ με την ε, ομάδα του, είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσουν εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να σας ακούσουν κυρίως. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαρνιέ για τη συμμετοχή σας, την παρουσία σας σήμερα εδώ και βεβαίως ε, και τον ηγετικό σας ρόλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πρωτοβουλία αυτή που θεωρούμε ότι αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για το πώς ε, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μπορούν να συνεργαστούν ε, για την προαγωγή των στόχων τους. Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στους εμπειρογνώμονες, Έχετε ακούσει τον Κρονέλη Διόγκα και φορέ φορές και σήμερα αυτή την εβδομάδα παρουσίασε μία από τις εκθέσει του. Θα του δώσω χρόνο ε, να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Μάλκολμ. Θα ξεκινήσω ομολογώντας το εξής. Ως ε, παιδί έπαιζα πολύ συχνά με ένα εικονικό ε, κατάστημα που είχα, τότε δεν υπήρχαν βιντεοπαιχνίδια και μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η ιδέα του να είμαι καταστηματάρχης, να πρέπει να ξέρω τι πρέπει να αγοράσω, τι γίνεται με τις τιμές. Όλη αυτή τη διαδικασία την έβλεπα, τη θεωρούσα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και από την άλλη έπρεπε να ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει τριγύρω μου, γιατί ξαφνικά υπήρχε μια επιδημία τριγύρω μου, ε, έπεφταν ε, οι τιμές ε, τρομερά και αν ο κόσμος δεν ήθελε ένα προϊόν, αλλά εγώ επέμενα να το έχω, τότε θα είχα σημαντικές ζημιές. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να παίρνει κανείς υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του καταναλωτή και του κοινωνικού ιστού. Γι' αυτό και ήταν πολύ ενδιαφέρον να εργαστώ για αυτή την ε, έκθεση παρακολούθησης ε, ε, μετά την έκθεση της Άννας Μαρίας για, την, για το λιανικό εμπόριο. Γιατί από οικονομικής πλευράς είναι βεβαίως εξαιρετικά σημαντικό. Γνωρίζουμε τα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη, το ΑΕΠ και την ανεργία. Ταυτόχρονα όμως έχει και τεράστιο κοινωνικό και πολιτιστικό αντίκτυπο το λιανεμπόριο. πλέον με την ολοένα και διευρυνόμενη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ε, έχουμε όλο και λιγότερες ε, δυνατότητες και ευκαιρίες ε, για κοινωνική συνάντηση. Και έτσι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και αυτή την αξία του λιανικού εμπορίου. Πέραν της οικονομικής υπάρχει και η κοινωνική πτυχή. Ιδίως πρέπει να αναδείξουμε και την αξία του μικρού καταστήματος που ε, αναλαμβάνει τεράστιους κινδύνους, ε, ιδίως μέσα στην κρίση, κάνει μια μεγάλη, δίνει μια μεγάλη μάχη, πρέπει να αναπτύξει ε, νέες ικανότητες με μια δραστηριότητα που είναι πολύ σημαντική για το χωριό, τη γειτονιά ή την πόλη. Επίσης εξέτασα τι έχει θέσει η Επιτροπή εντός αυτού του σχεδίου δράσης για το ελληνικό εμπόριο. Αυτό αφορούσε και η έκθεση εξάλλου. Η δική μου έκθεση ε, στηρίζει εν γέννη ε, τις ε, προτάσεις που αναφέρονται σε αυτό το σχέδιο δράσης. Υπάρχουν όμως δύο στοιχεία που δεν υπάρχουν και στην ΕΜΚΟ θα προσπαθήσουμε να, να συμπληρώσουμε το σχέδιο δράσης. Πολλοί λιανέμπορες μου έχουν πει ότι δεν υπάρχει πραγματική αναφορά ε, στην περίοδο που περνάμε, στην περίοδο κρίσης. Υπάρχουν ε, τόσα καταστήματα που κλείνουν, ε, χρεοκοπούν, την, τώρα τη στιγμή που μιλάμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν αυτό το στοιχείο και να δούμε πώς μπορούμε να αντισταθμίσουμε, αυτή την τάση, ότι δηλαδή τα καταστήματα κλείνουν. Επίσης, στο σχέδιο δράσης αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στον ανεξάρτητο λιανέμπορο και τη θέση του στην αγορά. Πώς ε, θα διασώσουμε τα παραδοσιακά καταστήματα, τα κέντρα των πόλεων για παράδειγμα. Στο σχέδιο δράσης τη Επιτροπής ε, δόθη ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να ε, προσέχουμε να μην πέσουμε στον προστατευτισμό βεβαίως. Από την άλλη όμως πρέπει να, τηρήσουμε, ε, να διατηρήσουμε και τα παραδοσιακά καταστήματα. Θέλουμε μικρά καταστήματα με ασφάλεια και ασφαλή κέντρα πόλεων. Ε, φτάνω και στο τέλος των πέντε ε, λεπτών μου. Το άλλο που ήθελα να θίξω είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές από μια άλλη οπτική γωνία, γιατί εδώ βλέπουμε την ε, συνεχή διαπάλη μεταξύ ε, των λιανεμπόρων και των ε, παραγωγών προμηθευτών. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Επίτροπος Μπανιέ προηγουμένως, ότι είναι καλύτερα να συνεργαζόμαστε με αυτή την αλληλοκατανόηση και γι' αυτό και στην έκθεσή μου δεν πρότεινα νέα νομοθεσία, γενικά το αποφεύγω. Ιδίως αφού υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες και εναλλακτικέ λύσεις. Έχω εντοπίσει όμως δύο αδυναμίες της εθελοντικής πρωτοβουλίας. Πρώτον, ε, για τους συμμετέχοντες θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρεία στήριξη και ισορροπία σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες και από την άλλη κάτι που ανέφερε και η Επιτροπή είναι το στοιχείο της επιβολής, της εφαρμογής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοια κρίση στις κάτω χώρες. Ξαφνικά τα σούπερ μάρκετ μπήκαν σε έναν πόλεμο τιμών που βεβαίως ε, είναι μια χαρά, δεν μπορώ να πω κάτι, ίσως να ωφελήσει και τους καταναλωτές γιατί πέφτουν οι τιμές. Από την άλλη όμω και κάποιε υπεραγορέ και σούπερ μάρκετ είπαν στου προμηθευτέ ότι εμεί δεν πρόκειται να απομισθούμε το κόστο ε, του πολέμου τιμών. Εσεί πρέπει να το κάνετε. Εσείς βρείτε τρόπο να μας δώσετε αυτά τα χρήματα, κυριολεκτικά, για να αντισταθμίσουμε αυτές τις, ε, τις απώλειες ε, του πολέμου τιμών. Αυτό βεβαίως είναι απαράδεκτο λαμβάνοντας υπόψη και τους κανόνες ε, της πρωτοβουλίας, της εθελοντικής πρωτοβουλίας. Ε, υπάρχουν σαφείς ε, πρακτικές, ε, όμως δεν εφαρμόζονται. Και τώρα βλέπουμε, είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται κάθε μέρα. Η κυβέρνηση των κατοχωρών θέλει να κάνει το διαμεσολαβητή μεταξύ προμηθευτών και υπεραγορών. Ξεκίνησε λοιπόν μια, ως μια εθελοντική πρωτοβουλία και τώρα στρέφονται προς την κυβέρνηση για να το λύσει. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο και γι' αυτό πρέπει να προσθέσουμε και κάποιες προειδοποιήσεις με το πνεύμα που ανέφερε και ο Επίτροπος Μπαρνιέ ότι είναι σημαντική και η υποβολή εφαρμογή πρέπει να βρούμε ε, κάποια άλλα μέτρα εάν η θελοντική πρωτοβουλία δεν είναι αποτελεσματική. Ευχαριστώ πολύ. Good. Ευχαριστούμε πολύ. Και την έκθεση αυτή θα την ψηφίσουμε ε, στο μέλλον, αλλά στα Χριστούγεννα. Απλώ τώρα κάναμε αυτή τη συζήτηση για να δοθεί και μια εικόνα. Εντάξει, τώρα θα περάσουμε ε, στον ε, πρώτον από τους ομιλητές μας, από το πάνελ μας, σε ό,τι φορά την άρση εμποδίων. Αυτό είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει αρχικά. Αυτή η στρογγυλή τράπεζα έχει ως στόχο να καταστήσει το ελληνικό εμπόριο πιο εύκολο, πιο αποτελεσματικό. Έτσι έχουμε αφήσει αρκετά ανοιχτή την ημερήσια διάταξη για να μας πούνε οι συμμετέχοντες σε ε, ποιες είναι οι λύσεις που προτείνουν. Ζερόμπερδιέ, θα πάρει πρώτα το λόγο. Ε, του ομίλου Καρφούρ. Και παλαιότερα έχει μιλήσει στο Κοινοβούλιο με άλλη ιδιότητα, μετά η κυρία Γκουνίλα Άνγκρεν της UEAPME, δεκεκριμένη οργάνωση ε, εκπροσώπησης των μικροψηφίων επιχειρήσεων εδώ στις Βρυξέλλες. Θα μας μιλήσει για τον ρόλο των μικροψηφίων επιχειρήσεων και τέλος, για πρώτη φορά νομίζω, υποδεχόμαστε τον Γκρέγορ ε, Βότσικ, ε, πρώην ε, CEO της Allegro στην Πολωνία, που ασχολείται κυρίως με το λιανεμπόριο στο διαδίκτυο. Και με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε πώς οι διαδικτυακές πωλήσει λαμβάνουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Θα σας δώσω 10 λεπτά στον καθένα. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε τις παρεμβάσεις σας και μετά θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους για ερωτήσεις παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Ο κύριος Μπεντιέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στα γαλλικά. Θα ήθελα καταρχάς εκ μέρους του ομίλου Καρφούρ να πω ότι Καλωσορίζουμε αυτή την πρωτοβουλία για τη συζήτηση του κυρίου Τραπέζης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Καρφούρ είναι όμιλος τοπικός και πολυμορφικός. Έχουμε πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ, αλλά και μικρότερα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, cash and carry, ηλεκτρονικό εμπόριο. Είμαστε τοπικοί, γιατί δρούμε σε διαφορετικά διαφορετικές, σε διαφορετικές περιοχές, σε περιφέρειες και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες πολλών διαφορετικών κοινωνιών με τα τοπικά τους γούστα και χαρακτηριστικά. 40% της, ε, του κύκλου εργασιών μας στη Γαλλία, δύο τρίτα συνολικά στην Ευρώπη. Πέρα της Γαλλίας είμαστε παρόντες στην, ε, στο Βέλγιο, την Ισπανία, τη Ρουμανία. Έχουμε franchising στην Ελλάδα. Και θα ήθελα, ξεκινώντας την ε, παρέμβασή μου, να μιλήσω για την απασχόληση. 360.000 συνεργάτες έχει ανά τον κόσμο ο Μίλος Καρφούρ πάνω από 200.000 στην Ευρώπη. Στη Γαλλία 110.000. Πρέπει να είμαστε ο πρώτος σε μέγεθος εργοδότης, ιδιώτης, στη Γαλλία. Και είμαστε πεπισμένοι ότι το μέλλον της επιχείρησής μας περνάει από την, από την εντατικοποίηση στην ε, απασχόληση. Διατηρούμε τις δραστηριότητες μας βέβαια και τα καταστήματά μας, εφόσον όμως αυτά μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες και έχουν το δυναμικό για ε, μια εμπειρία που θα προσφέρουν στον καταναλωτή και αυτό μπορούμε να το προσφέρουμε μόνο με ένταση απασχόλησης. Και αυτό πώς το κάνουμε, ανοίγουμε θέσεις για μαθητευομένους, ανοίγουμε ε, κρεοπολείο μέσα στα σούπερ μάρκετ μας και έτσι, αυτό είναι το κύριο μέλημά μας, να έχουμε δηλαδή ένα πλαίσιο λειτουργίας που θα επιτρέπει αυτή την, αυτόν τον εμπλουτισμό απασχόλησης διαφορετικά κινδυνεύουμε και πάλι να περάσουμε από το άχθος της παραγωγικότητας γιατί βέβαια αρκετοί προκειμένου να ε, εξηγήσουν ότι θα πρέπει να προσφέρουμε κάτι στην αγοραστική δύναμη μας έχουν επιβάλει, υποβάλει μάλλον σε μεγάλο άχθος παραγωγικότητας και εγώ θα ήθελα να περάσω σε λίγο σε μια επιχειρηματολογία ως προς την πίεση για όλο και χαμηλότερες τιμές που είναι παράλογη απέτηση. Και σε αυτό θα χρειαστούμε την υποστήριξη των δημοσίων κρατικών αρχών, γιατί αν οι δημόσιε αρχέ μα λένε συνέχεια ότι πρέπει και καλύτερα να πληρώνουμε τον παραγωγό και χαμηλότερε τιμέ να προσφέρουμε στον καταναλωτή, προφανώ δεν, δεν μπορούμε να ανθέξουμε αυτή την πίεση. Τι γίνεται λοιπόν για να αναπτύξουμε το εμπόριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα καταρχάς να υπογραμμίσω το πάρα πολύ σημαντικό έργο που έχει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά περισσότερο πρόσφατα, γίνει προκειμένου να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί η εσωτερική αγορά, μια συνεχής προσπάθεια, ένας αγώνας διαρκής που έχει αλλάξει πολλά πράγματα και που μας επιτρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη χωρίς πολλές δυσκολίες. Τούτου λεχθέντος όμως παραμένουν κάποια θέματα εκ των οποίων ορισμένα θα ήθελα να τα τονίσω πιο διεξοδικά προϊόντα λοιπόν θέματα φορολογίας και θέματα ρύθμισης του εμπορίου. Τα τρία θέματα στα οποία με τον τον άλλο τρόπο μπορεί να προκύψουν εμπόδια στις συναλλαγές. Για τα προϊόντα καταρχάς. Χρειάζεται λοιπόν διότι κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με μεγάλους προμηθευτές από, το, από τη διεθνή σκηνή, από τη διεθνή αγορά, ε, φυστάμεθα πολύ μεγάλες πιέσεις. Χρειαζόμαστε στήριξη λοιπόν σε αυτό, αλλά και σε τεχνικό επίπεδο υποστήριξη, γιατί έχουμε ζητήματα όσον αφορά τις, τους κανόνες για τα τρόφιμα που δεν είναι αρμονισμένοι, αλλά και νέοι κανόνες εμφανίζονται, όπως το Ρίτσεβι παραδείγματι, οι οποίοι δημιουργούν νέες προϋποθέσεις και απαιτήσει εναρμόνισης. Χρειαζόμαστε σε αυτό λοιπόν την δυνατότητα να διαχειριστούμε τις καταστάσεις με αποτελεσματικότητα. Αυτά για το προϊόν. δεύτερο θέμα για το προϊόν, η σήμανση, πολύ σημαντικό πιστεύουμε είναι... για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητα, η σήμανση προϊόντα όπως ε, το κρέας βιομηχανικής ε, παραγωγής. Αυτό που πρέπει να λέμε, πιστεύουμε πάνω στην ετικέτα, είναι όταν υπάρχει κατά 50% παρουσία ενός προϊόντος κρέατος, παραδείγμα τη λαζάνια με βοδινό κοιμά πάνω από 50% πρέπει να υπάρχει αναγραφή της προελεύσεως στην ετικέτα. Επίσης, οι Βρυξέλλες θα πρέπει να παρακολουθούν εάν γίνεται εναρμονισμένα η καταγραφή του Made in Germany, του Made in France, του Made in Italy. Πρέπει οι κανόνες που ισχύουν στην κάθε αγορά να είναι κοινοί, εναρμονισμένοι για να μπορούμε πιο δυναμικά να προχωρήσουμε στο ε, θέμα αυτό. Άλλο παράδειγμα. Οι μαζικές προσφυγές οι αγωγές που αποτελούν πιστεύω ε, κατάκτηση του καταναλωτή μεν, αλλά ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο στο κάθε κράτος και είναι ζητήματα που θα πρέπει να ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα περνάω στη φορολογία. Ως προς τη φορολογία έχουμε αφενός μεν θέματα διαφοροποιημένων συνθήκων ανάλογα με τη χώρα και έχουμε ένα πολύ γνωστό παράδειγμα. Στην Ισπανία επιβάλλεται φόρος σε καταστήματα ε, κάποιου μεγέθους, αλλά μόνο πάνω από κάποιο μέγεθος. Φόρος ο οποίος τελικά πλήττει τον αλλοδαπό περισσότερο από ότι τον εγχώριο καταστηματάρχη. Γιατί πληρώνουμε εμείς, σε παράδειγμα, 40% των φορών, ενώ καλύπτει μόνο το 8% της συνολικής επιφάνειας καταστημάτων στην Ισπανία. Να ένα παράδειγμα όπου υπάρχει <clears throat> ανάγκη για ε, ισότιμη αντιμετώπιση στη φορολογία. Άλλο παράδειγμα με τη φορολογία αυτό της πίστης σε σχέση ή της αφοσίωσης σε σχέση με το ε, διαδίκτυο. Ξέρετε ότι έχουμε φόρους διάφορους εγγύου ιδιοκτησίας ε, και άλλους πολλούς φόρους που έχουν να κάνουν με την συνήθιμα εμπορική δραστηριότητα. Από την άλλη όλοι έχουμε την, ε, τον αθέμητο ανταγωνισμό της πόλης μέσω του διαδικτύου που δεν υφίσταται την πίεση τη φορολογική και που επιπλέον επιβαρύνει και το εισόδημα της επιχείρησης με την ε, δυνατότητα εγκατάσταση σε διαφορετικά κράτη. Δηλαδή μπορεί να απαλλαγεί ακόμη και από το ΦΠΑ. Από ότι ο παραδοσιακό, θα έλεγα, καταστηματάρχη. Ξέρετε, αναγκάζομαι να χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό, γιατί ήμασταν κάποτε ο εξυγχρονισμό στο εμπόριο, αλλά τώρα πια ανήκουμε στην παράδοση. Φορολογία λοιπόν, ένα εκκρεμένο ζήτημα και οποιαδήποτε επιτεύγματα στον τομέα αυτό θα μας ε, είναι χρήσιμα. Η ρύθμιση των συναλλαγών, των εμπορικών συναλλαγών. Έχει προχωρήσει και στο θέμα αυτό η Ευρώπη, αφού έχει ληφθεί απόφαση για τις ε, αδειοδοτήσεις και την απαγόρευση της ε, επαλήθευσης οικονομικής ρόμης εν ανοίγματος καταστήματος. Τώρα λοιπόν μπορούμε να επαληθεύσουμε ή πρέπει να επαληθεύσουμε αν είναι εξίσου ανοιχτό ο τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξει σχετικέ ε, με τα εμπορικά καταστήματα και το εμπόριο γενικότερα. Επί παραδείγματι, οι ώρε λειτουργία καταστημάτων θα μπορούσαν να είναι μια λύση προκειμένου να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο, έτσι ώστε χωρί να θέλω να αμφισβητήσω βεβαίω ε, ε, η αδίποτε τοποθέτηση, να προδικάσω η αδίποτε πρόθεση των εργαζομένων, να μπορούμε να προσφέρουμε στον καταναλωτή μας ε, ώρες λειτουργίας καταστημάτων διαφορετικές και ασφαλώς ε, ευρύτερες από αυτές που γνώριζαν οι γονείς ή οι προπάποι μας. Και θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στην ανάγκη να υπάρχει ένα πλαίσιο ισορροπημένο σε σχέση με την άφηξη του ίντερνετ. Εμείς ξέρετε δεν έχουμε καμιά επιφύλαξη προς το ίντερνετ, άλλωστε ως όμιλος το αξιοποιούμε, το χρησιμοποιούμε, κάνουμε πολλή δουλειά και πολλές συναλλαγές χάρη στο ίντερνετ, ε, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε ε, ε, εξαιρετικές συνθήκες για το ίντερνετ και μεροληπτική αντιμετώπιση που μπορεί να, συμμετέχει, που μπορεί να συνεπάγεται ε, αθέμητο ανταγωνισμό. Επί παραδείγματο, όταν υπάρχει κάποιος ε, ε, μηχανισμό αναζήτηση, ε, μηχανή αναζήτηση, δεν μπορεί κανεί να τη χρησιμοποιεί δωρεάν προκειμένου να προβάλλει τη διαφήμιση του στον καταναλωτή απευθεία και δωρεάν. Μπορώ να συνεχίσω κύριε Πρόεδρε. Κάποια στοιχεία μόνο, πολύ σύντομα αν μου επιτρέπετε, που θα ήθελα να αναφέρω και που αποτελούν ένα, μια δυναμική θεώρηση, ένα δυναμικό όραμα που είναι τα ζητήματα της εγκύτητας, της εξέλιξης των πολεοδομικών ε, κέντρων, τα ζητήματα της τιμής ε, και βέβαια της ισορροπίας τιμής και ποιότητας ε, και πολλά άλλα ζητήματα που ευχαριστώ αν μου δώσετε το χρόνο θα επανέλθω και να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Αργότερα αν έχουμε χρόνο. Ούτως ή άλλως θα σας κάνουμε ερωτήσεις. Υπάρχουν διάφορα θέματα που ακούστηκαν. Επαναλαμβάνω, ε, μπορείτε να συμμετάσχετε μέσω του Twitter, αν θέλετε να συμμετάσχετε. Τώρα κυρία Αν Γκριν θα μας μιλήσει για την σκοπιά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, ως προμηθευτές. Ευχαριστώ, αγαπητοί φίλοι, βουλευτές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγχαίρω την Επιτροπή ΕΜΚΟ που οργανώνει την πρώτη ε, στρογγυλή τράπεζα για το λιανεμπόριο, γιατί αφορά έναν τομέα που είναι πολύ σημαντικός για τις ε, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ που εμείς που εκπροσωπούμε 12 εκατομμύρια ε, εργαζόμενους, μάλλον επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη, την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στη συζήτηση. Ε, στο πρόγραμμα γράφεται ότι είμαι εκπρόσωπος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δρούν ως ε, προμηθευτές. Σωστό είναι αυτό. Εγώ και ως ε, ιδιοκτήτης πολύ μικρής επιχείρησης ε, λειτουργώ και ως ε, προμηθευτής. Τα 30% των μελών μας είναι προμηθευτές. Μου να σχολιάσω το πώς μπορούμε να άρουμε τα εμπόδια, ούτως ώστε να υπάρχει ελευθερία της κίνησης, της εγκατάστασης και της επιλογής. Πριν ε, ξεκινήσω την παρουσίαση, θα πρέπει να τεθεί ένα προκαταρτικό και πιο σημαντικό ερώτημα. Δηλαδή, τι είδου ε, αγορά λιανεμπορίου θέλουμε στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολική να σας πω ότι μέχρι στιγμής δόθηκε πολύ μικρή προσοχή από την Ευρώπη στη δική μας κατάσταση των μικρών ανεξάρτητων ελιανεμπόρων. Επιπλέον, μερικές φορές παρουσιάζονται με πολύ αρνητικό, ας πούμε, με μια αρνητική απόχρωση. Τι σημαίνει λιανεμπόριο. Καταρχάς, πέρα από την, τις οικονομίες κλίμακας, για την, που είναι σημαντικό αυτό για την αποτελεσματικότητα, πρέπει να πούμε ότι εμείς ε, παρέχουμε πολλές ε, υπηρεσίες. Η οργάνωσή μου επί πολλά χρόνια θέλει να προωθήσουμε πρωτοβουλίες για να βελτιώσουμε τη λειτουργία της ε, εσωτερικής αγοράς. Μεγαλύτερη εναρμόνιση έχουμε ζητήσει, αλλά εναρμόνιση δεν σημαίνει κάτι την απόψή μας ότι δεν υπάρχει καμία ρύθμιση. Δεν μπορούμε να έχουμε ελεύθερο ανταγωνισμό χωρίς να εξασφαλίσουμε ότι η ελεύθερη αγορά υπάρχει, διορθώνονται οι ατέλειες και υπάρχει ισορροπία και δυνατότητα για κάθε παίκτη, μικρό ή μεγάλο, να έχει την ίδια ευκαιρία. Και ακριβώς αυτό συνέβη τα τελευταία χρόνια. Και αυτό ζητάνε μερικοί ακόμα. Να καταργηθούν οι εθνικές ρυθμίσεις που εξασφάλιζαν την ισοτιμία για όλους τους παίκτες, μικρούς και μεγάλους, του λιανεμπόριο. Στην ε, ΟΕΑΜΠΜΑ θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια ποικίλη αγορά όπου ο καταναλωτής μπορεί να επιλέγει ανάμεσα στις πολυεθνικές τις μικρές ε, φθηνές ε, αλυσίδες ή τα μικρά ανεξάρτητα τοπικά ε, μαγαζιά. Η εθνική νομοθεσία, οι εθνικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν την ισοτιμία για όλους. Παραδείγματο χάρη να μην πουλιάτε ένα προϊόν κάτω από το κόστος, γιατί αυτό σημαίνει όχι μόνο ε, δεχόμαστε τον, τον νόμο της ζούγκλας, αλλά και το δικαστήριο κατ' επανάληψη είπε ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτή η απαγόρευση. Επομένως, δεν πρέπει να ξαναμφιβητήσουμε αυτά τα πράγματα. Η δυνατότητα να διατηρήσουμε αυτή την απαγόρευση στις χώρες όπου υπάρχει είναι ζωτική σημασία για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ειδικά στον τομέα του λιανεμπορίου. Και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι αυτέ οι νομοθεσίε δεν είναι αποτελεσματικέ όπω ισχυρίζονται μερικοί. Ο στόχο αυτή τη νομοθεσία είναι να αποφύγουμε ότι οι μεγάλοι λιανέμποροι που πουλάνε με ζημιά έχουν κυρίαρχη θέση στην αγορά, πιέζουν συνεχεία τους μικρούς προμηθευτές για να αυξήσουν τις τιμές τους να δεχτούν μεγαλύτερε περιόδου αποπληρωμή, παραδείγματο χάρη 120 μέρε που έχω από μερικού πελάτες, να δεχτούν ε, πίστοση από κάποιους προμηθευτές. Ένα άλλο κρίσιμο θέμα είναι ε, οι κανόνες, οι αστικοί και οι τοπικοί. Η εγκύτητα των μαγαζιών ε, που δίνουν ε, ουσιαστικές ε, υπηρεσίες στους περίκους είναι πολύ σημαντικές για τους ηλικιωμένους αλλά και για τη ζωτικότητα πούμε, πόλεων, αεροκατοικημένων περιοχών κτλ. Από την οδηγία για τις υπηρεσίες δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο τα οικονομικά κριτήρια για την εγκατάσταση μιας επιχείρησης ή πιο συγκεκριμένα των σούπερ μάρκετ. Παρ' όλα αυτά η οργάνωσή μου πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να σέβονται τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα καταστήματα αυτά λιανεμπορίου είναι κυρίως ε, τοπικά μαγαζιά. Με βάση τα όσα πιστεύει η οργάνωσή μου, η Κομισιόν υπερεκτιμά το πώς αξοδεύουν οι καταναλωτές διασυνοριακά. Κάποιοι λόγοι για, που είναι το περιβάλλον, το αστικό περιβάλλον, η βιωσιμότητα των ε, κέντρων των πόλεων, η βιώσιμη κινητικότητα και η μεταφορά των αγαθών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τεθούν κάποιοι κανόνες για το άνοιγμα κάποιων καταστημάτων και να εξασφαλίσουν ε, ισοτιμία και ποικιλομορφία στην προσφορά. Θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε μελέτες που αναλύουν την επίπτωση των μεγάλων εμπορικών κέντρων ε, σε μια περιοχή. Λόγω των διαφορών στα κράτη-μέλη και διαφορετικών προσεγγίσεων που πρέπει να έχουμε, προκειμένου να λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση του κάθε κράτους μέλους, πολλά θέματα εξακολουθεί να πρέπει να τα αντιμετωπίσει το κράτος μέλος στο επίπεδό του. Αυτή η προσέγγιση έχει πλεονεκτήματα και είναι πολύ πιο σημαντική από την ε, λεγόμενη ε, άρση των εμποδίων που υπάρχουν στο διασυνοριακό ευρωπαϊκό εμπόριο. Φερρυπίν, οι κανονισμοί που αφορούν τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων ή θέματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα σε επίπεδο κρατών μελών δεν θα πρέπει να ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί μπορεί τότε όντως να υπάρχουν λιγότερα εμπόδια για διασυνοριακές συναλλαγές που είναι μια μειονότητα Αλλά όμως αυτά τα μέτρα πρέπει να προσαρμόζονται στις τοπικές ανάγκες στα κράτη-μέλη. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί κυρίες και κύριοι, οι μικροί λιανέμποροι θα πρέπει να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο. Πιστεύουμε ότι η φόρμουλα του franchise μπορεί να δώσει πολλά πλονεκτήματα για το λιανεμπόριο. Υπάρχει μεγάλη τάση μεταξύ των εταιριών franchise να επιβάλλουν ε, μία προμήθεια, ε, μία εγγύηση δηλαδή, για τους, στους λιανέμπορους. Ε, και αυτό ισχύει οριζόντια. Πιστεύουμε ότι οι μαζικές εξαιρέσεις στις κάθετες συμφωνίες θα πρέπει να αλλάξουν με τον εξή τρόπο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση να ανταγωνιστεί κανείς την περίοδο που ισχύει η σύμβαση. Ο κανονισμό θα έπρεπε να έχει μια διάταξη που θα λέει ότι οι μαζικέ εξαιρέσει δεν ισχύουν στι κάθετε συμφωνίε που περιέχουν μια ρήτρα όπου η αποτίμηση τη επιχείρηση καθορίζεται τη στιγμή της υπογραφή τη συμφωνία. Οι μαζικέ εξαιρέσει θα πρέπει επίση να μην ισχύουν εάν η συμφωνία έχει υποχρεώσει επιδόσεων που υποχρεώνουν τον αγοραστή να έχει ένα συγκεκριμένο κύκλο εργασιών με συγκεκριμένη περίοδο ή να αγοράσεις χι αριθμό αγαθών. Τέλος. Και για να σεβαστώ το χρόνο. Και αυτό θα ενδιαφέρει σίγουρα την ΙΜΚΟ. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι κάποιοι, κάποιες franchise προσπαθούν να προστατεύσουν τις αγορές τους ε, απέναντι σε ευρωπαϊκές ανταγωνιστικές ε, αλυσίδες. Εγώ τι προτείνω. Μια υποχρέωση ενός έτους ε, μη ανταγωνισμού, όπως αυτή που ανέφερα πριν, ή να εξασφαλίσουμε ότι οι όροι της σύμβασης δεν ανταποκρίνονται με την σύμβαση ενοικίασης, με τους όρους της σύμβασης ενοικίασης. Uh, well, thank you very much for some... Ευχαριστούμε πολύ. Έχω κάνει πολλές ε, σημειώσεις, ε, στις οποίες θα επανέλθω στη συνέχεια. Ξέρω ότι και ο Ντένις έχει κάνει πολλές ε, σημειώσεις γιατί αναφερθήκατε σε πολλά σημεία που καλύπτει στην έκθεσή του. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Gregory ε, Βότσεκ για να ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο πάνελ ομιλητών. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά ε, να βρίσκομαι εδώ με αυτή τη σύντομη ομιλία θα ήθελα να αναφερθώ ε, στα πιο σημαντικά ζητήματα. Τι πρέπει να καταλάβουμε για να ε, τονώσουμε την ε, οικονομία και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Μερικά εισαγωγικά σχόλια για να σας δείξω ποια είναι τα σημεία τα οποία θέλω να δείξω. Ουσιαστικά έχουμε δύο ε, δραστηριότητες, ο Όμιλος Αλέγκρο, ε, στον οποίο εργάστηκα για πολύ καιρό, και το e-Chamber, το ηλεκτρονικό επιμελητήριο που είναι μια νέα πρωτοβουλία στην Πολωνία, πριν από έξι μήνες ξεκίνησε, όπου διάφοροι ε, λιανέμποροι συνεργάζονται μέσω αυτού του ηλεκτρονικού επιμελητηρίου, κάνανε μια κοινή συζήτηση με εμπορευόμενους, και ε, εκπροσώπους των ε, υποδομών μέσω του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και της ε, επιστήμης της πληροφορικής. Ο Όμιλος Αλέγκρο είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ανατολική Ευρώπη, ξεκίνησε το 1999 και κινείται προς διαφορετικά τμήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, και αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται σε πάνω από 15 χώρες, ενέκ των οποίων είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απασχολούμε 6.500 Ευρωπαίους πολίτες. Θα αναφερθώ λοιπόν και σε, αυτή τη, σε αυτές τις διαφορετικές εμπειρίες ε, που είχαμε στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι όταν αναφερόμαστε σε ευκαιρίε στο εμπόριο, δεν μιλάμε μόνο για την εσωτερική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρούμε ότι είναι οικουμενική, παγκόσμια αυτή η ευκαιρία, γιατί δεν έχουμε θέσει εργασία και με το να τα κάνουμε όλα μόνο εσωτερικά δεν λύνουμε το πρόβλημά μα. Πρέπει να έχουμε και εσωτερική ανάπτυξη αλλά και εξαγωγέ. Στην Ευρώπη έχουμε πάνω από 250 εκατομμύρια ανθρώπους που ε, αγοράζουν προϊόντα στο διαδίκτυο. Αλλά πάνω από 530 εκατομμύρια ε, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, αλλά όχι για τις αγορές τους. Στην Ευρώπη είναι περίπου 35% το ε, ποσοστό των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Σε σχέση με άλλες ε, περιοχές του κόσμου δεν τα πάμε και άσχημα, αλλά και πάλι υπάρχουν ε, σημαντικά εμπόδια. Αυτή η ευκαιρία λοιπόν ανάπτυξης στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό επίπεδο θα πρέπει να βασιστεί ε, στην, ε, στην εμπορία υπηρεσιών εμπορευμάτων αλλά και υπηρεσιών. Και το τονίζω αυτό γιατί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία γιατί συνήθως τα ποσοστά, τα όρια κέρδους είναι μεγαλύτερα. Για Πάω στα πιο συγκεκριμένα τώρα. Το πρώτο και σκύριο αφορά τις δεξιότητες. Σε αυτό το νέο κόσμο πρέπει να δούμε ποιε είναι οι δεξιότητες που είναι σημαντικές. Ποιε θα μας βοηθήσουν να προοδεύσουμε. Και να άρουμε οποιοδήποτε εμπόδιο μπαίνει ανάμεσα σε εμά και σε αυτές τις δεξιότητες. Ε, ψηφιακή προσφορά, παρουσίαση του περιεχομένου, ε, τι θέλουμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές και στις άλλες επιχειρήσεις. Μετά, η εμπειρία του καταναλωτή ή του πελάτη. Γιατί είναι και ο τελικός ε, στόχος, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει η συναλλαγή. Για να τα καταφέρουμε, πρέπει να είναι όλο το οικοσύστημα μαζί. Πληρωμές, ε, τεχνικές πτυχές, αλλά και το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Όλες αυτές τις δεξιότητες. Ιδάλλως ε, δεν μπορούμε να πείσουμε τους πελάτες μας. Επομένως, αν θέλουμε μια δίκαιη και αναπτυσσόμενη αγορά πρέπει να σκεφτόμαστε όχι μόνο ε, βάσει των, των διαδικτυακών επιχειρήσεων, να σκεφτόμαστε ότι κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση είναι ηλεκτρονική επιχείρηση. Μπορεί να λέμε πάντα μία και ενιαία αγορά, πρέπει να λέμε πάντα να, να ακολουθούμε τους ε, τοπικούς καταναλωτές. Πιστέψτε με, Προσπαθήσαμε να ε, δημιουργήσουμε το ίδιο εμπορικό πρότυπο για μοντέλο σε πολλές διαφορετικές χώρες και πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι κανένα εμπορικό επιχειρηματικό μοντέλο δεν μπορεί να εφαρμοστεί ε, με τον ίδιο τρόπο ε, σε διαφορετικές χώρες. Πρέπει πάντα να προσαρμόζεται στα τοπικά δεδομένα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε και αυτό το online-offline γιατί είναι ένα στοιχείο προβληματισμού. Κάτι το οποίο πρέπει να ε, αναφέρουμε όμως εδώ ως πολύ σημαντικό είναι η κινητή τηλεφωνία. Ε, η IBM πέρσι έκανε μια μελέτη ε, για το από πού προκύπτει η ανάπτυξη και είπε το 3,7% προέρχεται από την εσωτερική κατάρτιση και 20% από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πολύ μεγαλύτερο λοιπόν το ποσοστό. Όταν όμως κατακαιρματίσαμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, βλέπουμε ότι πάνω από το 30% της ανάπτυξης προέρχεται από την κινητή τηλεφωνία. Επομένως, η αξιοποίηση αυτού του εργαλείου είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ του offline κόσμου, δηλαδή εκτός διαδικτύου, με ε, την διαδικτυακή εμπειρία. Και πραγματικά έχουμε πολύ καλά παραδείγματα στον τομέα. Για παράδειγμα, ε, ένας ε, κατασκευαστής χαλιών, ε, παραγωγός χαλιών με τεράστια λυσίδα καταστημάτων, αναφέρει ότι 50% των πελατών κάνουν έρευνα αγοράς πριν πάνε στο κατάστημα. Και αυτό είναι μια τρομερή ευκαιρία, γιατί ουσιαστικά έχουν συνδέσει τις υπηρεσίες που συνδέονται με, αυτή την, με αυτόν τον κλάδο και έτσι αύξησαν τα όρια κέρδους και ανάπτυξής τους. Όμως ε, υπάρχει και μια άλλη πτυχή. Δεν πρέπει να τα παίρνουμε όλα για δεδομένα. Πρέπει να ξεκινούμε από την αρχή, ε, να δοκιμάζουμε και να μαθαίνουμε. Να λαμβάνουμε υπόψη την, ε, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, την επιλογή των τιμών, διαθεσιμότητα, παροχή Ξέρω... Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει τρομερό ρυθμιστικό πλαίσιο στο διαδίκτυο θα ήθελα όμως να πω κάτι για τα, αυτά τα προσκόμματα. Πρέπει να άρουμε ε, τα προσκόμματα για την διασυνοριακή κατάρτιση. Οι υπηρεσίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια πλατφόρμα ανάπτυξης, αλλά και να υπάρξει και μια εξισορρόπηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Και θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ε, την ε, προστασία δεδομένων που να βασίζεται και να έχει ως κινητήριο μοχλό την ανάπτυξη. για αυτή την κατάρτιση πρέπει να δούμε ε, τι συμβαίνει με τα logistics, ε, την τεχνική πλευρά. Βεβαίως υπάρχουν ε, πολλά θετικά βήματα, αλλά μία από τις επιχειρήσεις που κατάφερε να μειώσει κατά 70% το κόστος των μεταφορών των δεμάτων έχει προβλήματα όμως γιατί οι αρχές μεταφορών λένε δεν έχει άδειε, πού είναι τα οχήματά σου. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια, ε, τέτοια παρανοϊκά <laughs> παραδείγματα. Και δεύτερον, πρέπει να είναι ε, με διπλή κατεύθυνση αυτή η παροχή υπηρεσιών αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να στείλει ένα δέμα από το Λονδίνο στην ε, Πράγα ή στη Βαρσοβία, αλλά το αντίστροφο κοστίζει τρεις φορές παραπάνω. Ενώ ακολουθείται η ίδια διαδρομή σχεδόν. Επίσης, δεν ξέρω πώς μπορεί να επιληθεί το ζήτημα του ΦΠΑ. Είναι σημαντικό. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε όμως με διάφορες ε, μεθόδους, εάν, κατα, αν υπάρχει δυνατότητα δραστηριοποίησης διασυνοριακά πιο εύκολα. Με τις ε, πλατφόρμες ε, υπηρεσιών πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα των πληρωμών, να υπάρχει ισότιμο πεδιοδογωνισμού. Γιατί ξέρουμε ότι πολλοί φορείς μπαίνουν πλέον στο παιχνίδι, τράπεζες και όχι μόνο, με, με τεράστιες δυνατότητες lobbying και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει θεμετό ανταγωνισμό. Και για το συμβατικό δίκαιο, Πολλέ φορέ το πρόβλημα υπάρχει με ε, τον ψηφιακό ή επιχάρτου μορφότυπο. Στον τουριστικό κλάδο βιομηχανία, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι μπορεί κάποιο να κλείσει ένα ξενοδοχείο, ένα ταξίδι, αλλά για να κλείσει όλε τι διακοπέ χρειάζεται να, έχει, ε, να τα τυπώσει όλα, γιατί ε, αυτό απαιτείται από το δίκαιο. στόχος ήταν να έχουμε μια, ένα τεκμηριωμένο μορφότυπο, αλλά όχι πάντα επί χάρτου. Για τα δικαιώματα των καταναλωτικών, λοιπόν, των καταναλωτών να έχουμε εναρμόνιση, αλλά όχι υπερβολικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι μικροψηφίε επιχειρήσει δεν θέλουν να προσπαθήσουν ε, την διασυνοριακή κατάρτιση, επειδή φοβούνται τον κίνδυνο οι πολιτικές επιστροφής θα πρέπει να ε, τηρούν και τα πρότυπα ε, καταπολέμησης της απάτης και ούτω καθεξής. Και τέλος, ε, για την προστασία δεδομένων, είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Με το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να έχουμε λύσεις που να μην σταματούν την καινοτομία, να έχουμε τέτοιες λύσεις που να προσαρμόζονται στην πραγματικότητα και να διατηρούμε και μια ευελιξία. Γιατί πάντα έχουμε τότε καλύτερα αποτελέσματα στην επαφή μας με τους, με τους ε, καταναλωτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Um, ευχαριστώ πολύ. Από το Twitter φαίνεται ότι ρωτάνε κάποιοι ποια είναι τα προσκόμματα στο διασυνοριακό εμπόριο. Μας τα καταγράψατε εσείς. Τα σημειώνουμε και σημειώνουμε και τα όσα λέτε για την προστασία που μπορεί να αποδείξει την ανάπτυξη. Έχουμε χρόνο για λίγες ερωτήσεις. Οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές, καταρχάς Χάιντι, Ντένις, Άννα Μαρία, Κυρία Ρούιλε, ευχαριστώ. Θα ήθελα από το τελευταίο ε, ομιλητή να ακούσω τι εννοεί ανάπτυξη με προστασία δεδομένων. Θέλετε, μιλώντα να λέτε και ποιοι είσαστε, γιατί εγώ μπορώ να σα γνωρίζω, αλλά δεν σα ξέρουν όλοι. Dennis Kredler από το European Retail Roundtable. Έχουμε ε, επιχειρήσεις λιανικής πόλης από 17 χώρες. Ευχαριστώ πολύ και για τελευταία παρέμβαση για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι η διάσταση αυτή όχι τόσο ορατή ακόμη. Στο λιανεμπόριο όμως έχει πολύ μεγάλο και πολύ ε, διαβροτικό χαρακτήρα, θα ανατρέψει τα πάντα ε, και δεν γνωρίζουμε καλά-καλά πώς θα εξελιχθεί το λιανικό εμπόριο με δεδομένο το ηλεκτρονικό. Όταν λοιπόν μιλούμε για φραγμούς στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ε, ασφαλώς θα πρέπει να δούμε και τους φραγμούς στο λιανεμπόριο. Ο συνάδελφος από το Αλέγκρο νωρίτερα μίλησε για φραγμούς στο εμπόριο πέραν των συνόρων. Βεβαίως συμφωνούμε με τον κατάλογο που ακούστηκε νωρίτερα, αλλά πολλές από τις, ε, πολλά από τα εμπόδια που αντιμετωπίσουν ε, οι επιχειρήσεις μας όταν θέλουν να ανοιχθούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο σε άλλες χώρες, κυρίως έχουν ε, να κάνουν με την μεταφορά του προϊόντος ή με ζητήματα σήμανσης και ενημέρωσης. Αυτό για να είμαστε απόλυτα σαφείς. Κύριο Χάρμπορ, δεν θέλουμε να μακρηγορείτε όμω, Κάντε μα την ερώτηση, σα παρακαλώ. Ευχαριστώ, ναι. Τα προσκόμματα αυτά πολλές φορές είναι έμεσο αποτέλεσμα νομοθεσιών και έχουμε καταθέσει μία πρόταση ε, με την ιδέα του, ε, της δοκιμής ηλεκτρονικού εμπορίου ε, και της αξιολόγησης των συνεπειών για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πιστεύετε ότι κάτι θα ήταν εφικτό. Ναι, ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, για να ακούσουμε και εσάς. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν έχω ερωτήσεις, κάποιες παρατηρήσεις μόνο, αλλά αν ακούτε ερωτήσει τότε θα περιμένω. Καλώς, όχι, θα σας πω λοιπόν τα εξή, ώστε το δυνατόν πιο σύντομο. Δύο παρατηρήσεις. Κριστιαν Βεσούρεν από το e Commerce μια ερώτηση για το round table και μια ερώτηση για τους ε, φραγμούς στην εσωτερική αγορά. Για το round table, για τη συζήτηση τρογγυλής είναι ευπρόσδεκτη η συζήτηση για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για την ενσωμάτωση της ιδέας του ηλεκτρονικού εμπορίου σε κάθε ε, υιοθετούμενη νέα νομοθεσία και ίσως θα πρέπει στο εγγύς μέλλον ένα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα να κοιτάξει τη, μεγάλη ποικιλία μέσων που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Υπάρχουν πάρα πολλά μέσα, πάρα πολλοί φορείς και πάρα πολλές υπηρεσίες και προϊόντα. Ε, ωστόσο, εκπροσώπους καταναλωτών δεν έχουμε στον τομέα αυτών και πολύ ευχαριστώ να σας υποστηρίξουμε με τον ε, χρόνο που έχουμε στη θέση μας εδώ. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ε, αγορά λιανικού εμπορίου και δεν πρέπει να λησμονούμε την αγορά όταν συζητούμε εδώ. Οι επιχείρησεις, οι θέσεις εργασίας προσφέρουν αυτές, οι οποίες είναι πάντα εγχώριες, τοπικού χαρακτήρα, δεν προέρχονται από έξω ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές και σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε σε μια δύσκολη περίοδο, όπως άλλωστε είχε γίνει και το 2004 με τη μεγάλη ε, διεύρυνση όπου οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και όχι μόνο διεθνούς χαρακτήρα, ανασκουμπόθηκαν για να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις πάνω από 100 και 400 400.000 εργασίας. Εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι μπορούν ε, οι, καταστα... οι επιχειρηματίες επιχειρήσεις ελληνικού εμπορίου να πηθήσουν και στην αγορά εργασίας. Και ως προς τα εμπόδια που ακούστηκαν νωρίτερα από τον κύριο Μπεντιέ για τη φορολογία, ε, για τις ε, δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά και όλα αυτά, θέλουμε να τα υπογραμμίσουμε. Η κυρία Μπίλτ αλλά και ο κύριος Φαπ πιστεύω θα πρέπει να κοιτάξουν προσεκτικά τις αρχές της ιστορικής αγοράς, τις αμοιβές αναγνώρισης και θα σας παρακαλούσαμε να επικεντρωθείτε σε αυτές. Όπως είπα από την αρχή Ανα Μαρία, ο στόχος αυτής της συζήτησης του Ικλής Τραπέζης ήταν ακριβώς να ακουστούν όλων οι φωνές. Μια πρώτη απόπειρα είναι. Πολύ ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας και ακούμε τον επόμενο μιλητή. Εσείς πρώτα και μετά ο άλλος, ναι, ευχαριστώ πρόεδρε, λέγομαι Λέρνεκερ, εκ μέρου της ΕΔΙΚΟ, που είναι μια συνεταιριστική οργάνωση επιχειρηματιών λιανικής, λιανικών πωλήσεων που έχει κύκλο περίπου 45 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Το θέμα του κόστους. Ε, μην Ε, επιμένετε και κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις πωλήσει κάτω του κόστους. Απορρίπτουμε πλήρως αυτή την ε, ε, πρόταση. Έχουμε καταρχάς τις αρχές μονοπωλίου και ανταγωνισμού της Γερμανίας, οι οποίες λένε ότι δεν υπάρχει βάση για τέτοιου τους απαγόρευση. Επίσης όλα τα νομικά περιοδικά η θεωρία νομική και όλοι οι καθηγητές θεωρούν ότι ακριβώς αυτό συμβαίνει, δηλαδή οι οικονομικές συνέπειες δεν είναι πάρα πολύ χαμηλές και εν τέλει η οικουμενική ε, δικαιοδοσία του γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου θα κατηθιστούσε μια τέτοια διάταξη μη εφαρμόσιμη, λέει στα αγγλικά ο ομιλητής θα σας παρακαλούσα να το λάβετε υπόψη. Η απαγόρευση αυτή είναι απολύτως άχρηστη. Ο κύριος Χάρπορ. Από το 99 που έρθα στο κοινοβούλιο είχαμε μια πρόταση από την Επιτροπή για την πρόθεση των πολίσεων, η οποία είχε και μεταξύ αποσυρθεί, αν δεν αποτώνα. Με πολλά επιχειρήματα υπέρ της απαγόρευσης στην Ευρώπη των πωλήσεων κάτω του κόστου κτλ. Αλλά δεν το υποστήριξαν όλα τα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι ένα από τα θέματα που πρέπει να παραμένει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών όσο ζήτημα επικουρικότητα είναι αυτό. Αλλά ήταν ενδιαφέρουσα η παρατήρηση σας. Η κυρία εκεί στο κέντρο πίσω και ίσως και κάποιος άλλος έχει στήσει το λόγο. Με τις δύο αυτές παρεμβάσεις λοιπόν θα κλείσει αυτός ο γύρος συζητήσεων και θα δώσω και στους ομιλητές μας στο τέλος ένα λεπτό στον καθέναν για να δώσουν σύντομα κάποιες απαντήσεις αν έχουν. Χωρίς μικρόφωνο. Μίριαμ Φαντεστίχελε από το Άμστερνταμ. Έχω μια ερώτηση για την δοκιμή οικονομικών αναγκών. Φαίνεται ότι Υπάρχει ανάγκη για εφαρμογή της για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών. Οι υπηρεσίες λοιπόν και οι συμφωνίες για το ελεύθερο εμπόριο που συνεχίζουμε να, που συνάπτουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν κάποια εφαρμογή εδώ. Επίσης θέλω να πω ότι αναφέρεται με μεγάλη ικανοποίηση η κατάργηση της υποχρέωσης δοκιμής ε, αποτελεσμάτων. Αλλά αυτό έρχεται σε αντίφαση με την ε, έκθεση του κυρίου Νταγιόγκ. Μπορεί κανείς να μας εξηγήσει πώς μπορεί να γίνει πιο ευέλικτη αυτή η δοκιμή οικονομικών αναγκών. Πώς οι εθελοντικές πρωτοβουλίες, ρώτησε κάποιος, μπορεί να δουλέψουν χωρίς ε, εμπιστοσύνη τέθηκε αυτό το ερώτημα στο Twitter, στο ίντερνετ. Η κυρία εκεί με τα καφέ, με το μικρόφωνο σας, από την Οργάνωση Ανεξάρτητων Λιανεμπόρων. Τρία σύντομα σχόλια. Πρώτον, μου άρεσε αυτό που είπε ο κύριος Ντε για την πυκλομορφία της ευρωπαϊκής αγοράς και τους πολυπίκυλους φορείς που δραστηριοποιούνται, αυτή η ποικιλομορφία συχνά θεωρείται δεδομένη από τους καταναλωτές ή την αγνοούν. Ε, μεγάλη, έχουμε μεγάλη πλειοψηφία ε, μεγάλων υπερκαταστημάτων αλλά και ανεξάρτητων μικρών λιανεμπόρων. Ε, με αυτόν τον τρόπο έχουμε ανεξάρτητη βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Χαίρομαι λοιπόν όπου αυτή η μοναδική πτυχή της αγοράς μας ε, υποστηρίζεται από αυτή την έκθεση. Το αν κρατήσουμε αυτή την πυκλομορφία και την προωθήσουμε σε όλα τα κράτη-μέλη είναι πολύ σημαντικό. Το να προωθήσουμε την πυκλομορφία και την νοοτροπία την επιχειρηματική είναι πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά για τις ανατολικές, ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες όπου είναι υπανάπτυκτες ακόμη αγορές και έχουν λιγότερη ποικιλομορφία. Ε, κύριε De Young, να προσθέσουμε ε, δύο πράγματα. Η θέση των εξάρτητων λιανεμπόρων και το κλείσμα των καταστημάτων. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα μπορεί να, προσφέρουν λύσεις, αξίζει να τις διερευνήσουμε. Ε, καλό θα ήταν, ε, αν θέλετε, περιπτώσει, να σας εξηγήσω τα διάφορα μοντέλα στα οποία πιστεύω. Ευχαριστώ για αυτές τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλο θέλει να ξαναπάρει το λόγο. Να δώσω το λόγο καταρχάς στον Ζερόμ Μπιντιέ μπορείτε να σχολιάσετε, να απαντήσετε σε οποιαδήποτε από τα ερωτήματα ακούσατε. Να διαλέξετε δηλαδή τις απαντήσεις και πού θα απαντήσετε. Για τα θέματα της ρύθμισης των σχέσεων με τους προμηθευτές και τα θέματα των αγορών. Συμφωνούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν πωλήσει κάτω από το κόστος και είμαστε γενικά αντίθετοι ε, βεβαίως και στις τιμές της ε, ληστρικές. Η πεποίθησή μας είναι ότι θα πρέπει να βγούμε από αυτή την ε, ατμόσφαιρα ε, προβολής του χαμηλού κόστους, όπου συστηματικά προτάσετε το χαμηλό κόστος, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας προσφέροντας μια πλειάδα προϊόντων χάρη σε μόνιμες, μεσοπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους, ε, μακροπρόθεσμες επαφές με τους προμηθευτές μας. Έχουμε διάφορα προϊόντα, έχουμε γεωργικά προϊόντα, ε, για τα οποία έχουμε συμβάσεις με τους γεωργούς και που παραμένουν αυτοί οι γεωργοί προμηθευτές μας για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να βγούμε από αυτή τη συζήτηση πια του low cost, του χαμηλού κόστους. Ήταν πάρα πολύ σκληρή αυτή η θεωρία για τον τομέα μας ε, και που αναπτύχθηκε ειδικά πάρα πολύ με το ίντερνετ και είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο να προωθήσει ένα εμπόριο που θα δημιουργεί αξίες. Καταρχάς για μας ε, η καρδιά των εμπορικών σχέσεων είναι ο σεβασμός της σύμβασης, της, της συμφωνίας, της σύμβασης δηλαδή. Κύριε, όπως είπε και ο κύριος Μπαρνιέ, πιστεύουμε πολύ περισσότερο στη σύμβαση παρά στις ρυθμίσεις. Καλό είναι να έχουμε καλές συμβάσεις, παρά να έχουμε μετά νομοθετικά κείμενα. Πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να γίνονται σεβαστές οι συμβάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να μπορούμε να δουλεύουμε. Τρίτο ερώτημα. Στη σχέση μας με τους προμηθευτές θα ήταν πολύ επικίνδυνο να μπερδέψουμε και να βάλουμε τους πάντες. Γιατί πριν από εμά υπάρχουν πάρα πολλοί ε, φορείς. Έχουμε μεγάλες πολυεθνικές που έχουν τεράστια εμπορική δύναμη. Και συχνά μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντική αυτή η δύναμή τους από εμά. Έχουμε συνεχεία μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις οποίες πρέπει να έχουμε ειδικά συστήματα διαλόγου και φυσικά θέλουμε να τα κρατήσουμε και βεβαίως έχουμε και τους ε, γεωργούς από τους οποίους δεν αγοράζουμε απευθείας. Ε, συνήθως αγοράζουμε από βιομηχανικές εταιρείες, όχι απευθείας από τους γεωργούς. Θα πρέπει λοιπόν στις σχέσεις αυτές εμπορίου βιομηχανίας να λάβουμε υπόψη μας τις διαφορετικές αυτές σχέσεις. Ε, τώρα, εμείς εντασσόμαστε σε αυτή τη λογική του action plan, του σχεδίου α, δράσης που λαμβάνει υπόψη μας τις δυνατότητες να δημιουργήσουμε ζώνες όπου αναμειγνύεται το εμπόριο ε, με άλλες δραστηριότητε και βεβαίως ε, λαμβάνει υπόψη και η διάσταση του περιβάλλοντος. Σε όλα αυτά θέλουμε να παίξουμε το ρόλο μας. Ευχαριστώ, λέει κυρία Αλμγκρεν. Τι μπορώ να πω εγώ ως επιχειρηματίας και ίδια. Για μας τους επιχειρηματίες είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε κυρίως για τους ανεξάρτητους ε, επιχειρηματίες. Σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις δεν έχετε ποτέ πραγματογνωμοσύνη, δεν έχετε ποτέ ειδικού. Συχνά ο καθένας είναι μόνος του. Ε, αντιμέτωπος με την νομοθεσία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να είναι εύληπτη η νομοθεσία, να μπορούμε να τη βρούμε εύκολα. Και βεβαίως θα πρέπει οι εθνικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι είναι σταθερές οι ρυθμίσεις, να μην αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο. Και βεβαίως αυτό που περιμένουμε με αδημονία είναι ότι πρέπει να λαμβάνετε, περιμένουμε να δούμε στην πράξη να εφαρμόζεται η αρχή του Think Small First. Έχουμε δηλαδή πρώτο μας μέλημα και πρώτη μας ε, μέρημνα τις μικρές επιχειρήσεις για τις ε, ρυθμίσεις. Να πω κάτι σημαντικό, ένα σημαντικό πόρισμα. Κάναμε ένα ερωτηματολόγιο ε, και το απευθύναμε σε διάφορους ε, φορείς για τη νέα οδηγία για τους καταναλωτές. Και αυτό που είναι περίεργο ήταν ότι το αποτέλεσμα, αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μάλλον στο ερωτηματολόγιο είπαν, πέστε μας δύο εβδομάδες πριν, όταν εφαρμοστεί, εμείς τι πρέπει να αλλάξουμε στην ιστοσελίδα. Έτσι αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει την νομοθεσία. Δεν μπορούν, δεν έχουν πόρου να παρακολουθήσουν την νομοθεσία. Μην πω ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να υποφεληθούν από αυτήν. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Είναι πολύ σημαντικό. Και όταν μιλάω για ανάπτυξη, σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάμε κάθε είδους νομοθεσία πώς την ερμηνεύουν, πώς την αντιλαμβάνονται εκείνοι που δεν έχουν στρατιές δικηγόρων από πίσω να τους την εξηγούν. Θα πρέπει να είναι εύκολη να εφαρμοστεί. Και μόνο τότε έχει αξία. Μοιάζει απλοϊκό αυτό που λέω, αλλά όταν δείτε οποιοδήποτε κείμενο, με αυτό το κριτήριο θα καταλάβετε πόσο περίπλοκα είναι αυτά τα κείμενα. Τι θέλω να σας πω λοιπόν. Εντάξει, εναρμόνιση. Καλή είναι, απαραίτητη είναι, οπωσδήποτε. Πρέπει πάντα να ακολουθούμε τις συνήθειες των καταναλωτών, γιατί δεν είναι εύκολο να τσαλάξουμε αυτές τις συνήθειες, πρέπει να τις καταλάβουμε και να αντιδράσουμε. Αλλά όχι υπερβολικά πολλές ρυθμίσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θέλουν να εξάγουν γιατί αντιμετωπίζουν τεράστιο ρίσκο. Ήδη ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι τεράστιος. Στην Ευρωζώνη δεν το αισθάνεστε πολύ αυτό, αλλά μην ξεχνάτε ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης δεν είναι Ευρωζώνη και οι εξαγωγές ανέχουν αυτόν τον κίνδυνο του συναλλάγματος. Επίσης, τι γίνεται με την ροή χρήματος. Τώρα για την προστασία των δεδομένων με ανάπτυξη. Προσοχή λοιπόν, πού πρέπει να προστατεύσουμε δεδομένα και πότε. Να μην σταματήσετε την καινοτομία, όμως, αλλά όλα αυτά να τα βάζετε στο σωστό πλαίσιο, να έχετε τους ορισμούς σας απλούς, εύληπτους σε όλα τα νομοθετικά κείμενα. Αυτά. Αυτά ε, ήταν οι σκέψεις που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ευχαριστούμε. Βεβαίω θα πρέπει να απευθύνουμε αυτά τα σχόλια και στου συναδέλφου από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να δούμε και τι δικέ του παρατηρήσει. Σα περάσουμε τώρα στο δεύτερο πάνελ με του επόμενου ομιλητέ, του οποίου καλωσορίζω. Όπω ε, ανέφερα προηγουμένω, το δεύτερο στοιχείο θα αφορά την ευθύνη και την ε, ισότητα Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσουμε τον κύριο Ροντρίγκο Κουβέια, Γενικό Γραμματέα ε, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ε, Καταναλωτών, της Eurocoop. Προέρχεται την Πορτογαλία, με μεγάλη εμπειρία σε αυτό το τομέα. Και μετά θα, θα συζητήσουμε και το θέμα της ε, αγοράς του purchasing με τον Jean-Denis Deveyna από την Auchan άλλη μια μεγάλη γαλλική εταιρεία λιανεμπορίου και με μεγάλη χαρά για πρώτη φορά στην Επιτροπή μας, παρότι πολλές φορές συμμετέχει στην Επιτροπή Άγκρη, καλώς με τον κύριο Πέκα Πέσονεν. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ. Γενικός Γραμματέας της Κόπα Κοτζέκα το γεωργικό λόμπι που εκπροσωπεί 70% των οργανώσεων παραγωγών στην ε, Ευρώπη. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κουβέλια για να μας δώσει τη δική του οπτική και μετά συνεχίζουμε. Έχετε 10 λεπτά. Thank you, Chairman. Uh, thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν θα μιλήσουμε την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα της UCOP ε, αλλά ως ε, συμπρόεδρος ε, της ομάδας διαχείρισης ε, της πρωτοβουλίας συγγνώμη, της πρωτοβουλίας για την αλυσίδα εφοδιασμού. Όπως τη γνωρίζετε εσείς, μάλλον θα είναι εθελοντική πρωτοβουλία. Η επίσημη ονομασία είναι Supply Chain Initiative, όπως βλέπετε και στην οθόνη σας. Θα περιγράψω εν συντομία τι έχουμε κάνει, τι έχουμε επιτύχει έως τώρα και πώς θα που κάτι που θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Ξεκινήσαμε με τη συζήτηση για τις ε, αρχές ε, των ε, θεμητών εμπορικών πρακτικών και αυτό αφορά όλους τους φορείς από τους γεωργούς, στους μεταποιητές, στις μικρότερες επιχειρήσεις, λιανεμπόρους και τον Νοέμβριο του 2011 καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα σύνολο 10 αρχών που αφορούν την δικαιοσύνη των εισαγωγικών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Υπάρχουν τρεις γενικές και εφτά πιο ειδικέ αρχές. Δεν θα εξέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Βεβαίως, πέραν αυτών των αρχών, αναγνωρίστηκε ότι η συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο συμπεριλαμβανομένου και του δίκαιου ανταγωνισμού είναι μια πολύ σημαντική πτυχή. Μαζί με αυτές τις αρχές επίσης ε, καταλήξαμε σε παραδείγματα θεμητών και αθέμητων πρακτικών κατά τη γνώμη μας για κάποια πολύ συγκεκριμένα ζητήματα όπως ε, οι ε, γραπτές ή προφορικές συμφωνίες, γενικοί όροι και προϋποθέσεις και ούτω καθεξής. όλες αυτές οι οργανώσεις ε, στο σύνολο της τροφικής αλυσίδας συμφώνησαν από αυτών των παραδειγμάτων. Έγιναν θερμά υποδεκτά όλα αυτά από το ε, Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου της Επιτροπής για την ε, Εποπτεία της Τροφικής Αλυσίδας που μας ζήτησε στη συνέχεια να αναπτύξουμε ένα πλαίσιο για την εφαρμογή και επιβολή αυτών των αρχών. Αυτό κάναμε λοιπόν στη συνέχεια. Ξεκινήσαμε το διάλογο και τον Ιανουάριο 2013, φέτος δηλαδή, καταλήξαμε σε ένα πλαίσιο για την εφαρμογή των αρχών. Δυστυχώς, εκείνη την περίοδο δεν ε, κατοχυρώσαμε τη σύμφωνη γνώμη όλων των εταίρων ε, στη συζήτηση, ιδίως της ΚΟΠΚΟΖΕΚ που εκπροσωπούσε τους γεωργούς και τη τράβη που εκπροσωπούσε τους μεταποιητές κρέατος. Ε, παρότι η έτερη ε, συμμετείχε στην Food King Europe και έτσι μπορεί να θεωρηθεί ότι συμφωνούν και συμμετέχουν ε, στη συμφωνία μέσω της οργάνωσης τροφίμων και ποτών Ευρώπης. Αυτό το πλαίσιο έχει δύο πτυχές. Αφενός εστιάζεται στην πρόληψη. Πώς δηλαδή διασφαλίζουμε ότι οι αθέμητες ε, πρακτικές δεν ε, χρησιμοποιούνται στην αγορά ή ακόμα καλύτερα πώς ε, θα διασφαλίσουμε ότι θα ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις πάντα οι θεμητές πρακτικές. Τουλάχιστον από τις εταιρείε που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μας. Πρόληψη λοιπόν πρώτον. Δεύτερον, τα 11 μέσα. Τι συμβαίνει δηλαδή όταν αυτές οι πρακτικές ε, δεν συνάδουν με τις αρχές που έχουμε θέσει. Πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα. Έχουμε εδώ κάποια, κάποιες δεσμεύσεις, αφενός ε, βεβαίως να, γίνουν, να σεβαστούν επιχειρήσεις στις αρχές και δεύτερη δέσμευση να σέβονται και τη διαδικασία. Αυτό το εγχείρημα εποπτεύεται από ε, μια ομάδα διακυβέρνησης, της οποίας συμπροεδρεύω από πλευράς ελληνικού εμπορίου και ο συμπρόεδρος μου, η συμπρόεδρος μου Χόξαν Φιλέρ είναι συμπρόεδρος από πλευράς βιομηχανίας. Είναι Διευθύντρια ε, στην ε, Ένωση Τροφίμων και Ποδών Ευρώπης και βεβαίως έχουμε και εκπροσώπους από την ε, τροφική αλυσίδα, λιανικό εμπόριο και χονδρεμπόριο. Δυστυχώς οι γεωργοί δεν εκπροσωπούνται ακόμα, όπως ανέφερα και προηγουμένως, αλλά συνεχίζουμε το διάλογο. Έχουν προσκληθεί ως παρατηρητές Βρισκόμαστε σε συζητήσεις και ελπίζουμε στο προσεχές μέλλον ε, να καταφέρουμε να οικοδομήσουμε αυτή τη γέφυρα που θα μας επιτρέψει να κινηθούμε εκ παραλίλου στο μέλλον. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, δεν έχω χρόνο. Ουσιαστικά όμως η ομάδα διακυβέρνησης βασίζεται στη συνένεση, έχει κανόνες εμπιστευτικότητας ε, σε ό,τι αφορά τις ε, συζητήσεις σε ορισμένε περιπτώσει υπάρχει και ένας βαθμός ανωνυμία και βεβαίως νομική συμμόρφωση, προφανώς. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε συμπεριλάβει ε, και μια ειδική περίπτωση ε, όπου αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις ε, όπου θεμι, μη θεμητές ε, πρακτικές συσσωρευμένης διαφοράς, ας πούμε, όταν μια θέμητη πρακτική επηρεάζει μια ομάδα επιχειρηματιών, οι οποίοι κινούνται από κοινού, αν δεν υπάρχει μια πλατφόρμα στο εθνικό επίπεδο ή υπάρχει μεθοριακή διάσταση, το η ομάδα διακυβέρνηση αυτή, το Governance Group, θα χειριστεί την υπόθεση για να δώσει κατευθυντήριε γραμμές για τη διευθέτηση των διαφορών. Έχουμε αναπτύξει και κάποια εργαλεία για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές. Ένα μέσο αυτοεξιολόγησης για να ελέγχουν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ε, σε σχέση με τις αρχές μας και πώς μπορούν να βελτιωθούν. Έχουμε ένα εργαλείο ηλεκτρονικής εκμάθησης, e-learning, που θα βοηθήσει ε, το προσωπικό της επιχείρησης να καταρτιστεί. Υπάρχουν κάποιες γλωσσικές εκδοχές, ε, αναπτύσσονται και άλλες μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου και αν επιθυμείτε να έχετε και γλώσσες μπορείτε να μας το πείτε. Βλέπετε στην οθόνη τον ιστότοπο. Έχουμε όλη την φιλοσοφία μας ε, εκεί, η οποία περιγράφεται αναλυτικά. Μπορείτε να γραφτείτε ε, στο ιστότοπό μας και ε, αναφέρονται και οι εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μας. Και με τα χαράς μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει επιστολές ενδιαφέροντος από πάνω από 80 επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη που εκπροσωπούν στις εθνικές αγορές πάνω από 450 ε, εταιρείες. Οι μισές από αυτές είναι τοπικές και άλλες, υπάρχουν και μεγάλες πολυεθνικές και είπαν ότι όταν θα είναι απολύτως έτοιμες θα εγγραφούν και εκείνες στην ε, εθελοντική πρωτοβουλία της τροφικής αλυσίδας. Βεβαίως υπάρχουν ε, μεγάλες πολυεθνικές ε, λιανικού εμπορίου, υπάρχουν μεταποιητές, υπάρχουν συνεταιρισμοί, ανεξάρτητοι ε, λιανέμποροι, υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Θα ήθελα να πω ότι αυτές οι επιχειρήσεις εκπροσωπούν ουσιαστικά χιλιάδες ε, εμπορικούς εταίρους. Όταν ξεκινήσουν λοιπόν να εφαρμόζουν ε, ε, αυτές τις αρχές, αυτό θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και έτσι θα επηρεάσουν πολλές πολλές ακόμα επιχειρήσεις στην Ευρώπη και έτσι αυτές οι εταιρείε μικρού μεσαίου μεγέθους, οι γεωργοί, οι μεγάλες επιχειρήσεις όλοι θα επωφεληθούν από την εφαρμογή αυτών των ε, βέλτιστων πρακτικών. Έτσι ξεπερνάμε ακόμα και τις δικές μας ε, προσδοκίες. Ε, τελειώνει ο χρόνος μου βλέπω, οπότε κλείνοντας να πω ποια είναι τα βήματά μας για το μέλλον. Ξέρουμε ότι η κατάσταση δεν είναι ιδανική, αλλιώς δεν θα υπήρχε και λόγος να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Όμως η ουσία είναι ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να δείξουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα της αγοράς. Και δεν πρέπει να κρίνουμε την αγορά, ε, την πρωτοβουλία, συγγνώμη, βάση παραδειγμάτων του παρελθόντος, γιατί ξεκίνησε επισήμως στις 16 Σεπτεμβρίου. Πρέπει λοιπόν να κοιτάζουμε προς το μέλλον και να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Βρισκόμαστε στην αρχή για να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με τα ε, προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Είμαστε πεπισμένοι, ξέρουμε μάλλον ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ζητήματα, είμαστε όμως και πεπισμένοι ότι έχουμε τη λύση. Χρειαζόμαστε χρόνο για να δείξουμε ότι αυτή είναι η πραγματική λύση των προβλημάτων μας και ελπίζουμε τα ευρωπαϊκά όργανα να μας στηρίξουν. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ. Συγγνώμη, δεν σα ανέφερα μεγαλύτερα. Σε βλέπω, ότι με χαρά, βλέπω με χαρά ότι έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. οποίο ενδιαφέρεται μπορεί και από το διαδίκτυο να πάρει τι πληροφορίες και να στείλει τα μηνύματά του μέσα του Twitter. Και τώρα, παρακαλώ τον κύριο Ντεβάινε να μας μιλήσει. Έχετε μεγάλη εμπειρία από το Ιουλιανικό Εμπόριο και τον Όμιλο Οσό. Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση που δείχνει πόσο σημαντικό ρόλο σκοπεύει να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια αλυσίδα λιανικού εμπορίου πιο αποτελεσματική και πιο ισότιμη. Θα μιλήσω όμως πρώτα για τον Όμιλο Οσό. Γαλλικό όμιλο Νανικού Εμπορίου παρόντα σε 13 ευρωπαϊκά κράτη, εκ των οποίων 8 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κύρια δραστηριότητα το υπερ σούπερ μάρκετ, το πολύ μεγάλο, 800 έχουμε, 3.000 σούπερ μάρκετ απλά και πολλά επίσης ε, ε, εμπορικά κέντρα. Μας ενδιαφέρει πολύ το ε, ηλεκτρονικό εμπόριο, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που εφήβραμε τον drive στη Γαλλία. Και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στον τρόπο με τον οποίο ο μιλός μας αντιλαμβάνεται τις εμπορικές συναλλαγές και κυρίως τις σχέσεις τους με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφενός, αφετέρου τις ε, ε, ανάγκες που έχουν ξεπεράσει τα παραδοσιακά όρια σε σχέση με την ε, διαπραγμάτευση και την ε, θέση των διαπραγματευομένων και τρίτον να πω γιατί θεωρώ, θεωρούμε ως ομιλοσουσό ότι μια κανονιστική προσέγγιση δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα. Για να, κατα... για να φτιάξουμε λοιπόν τις σχέσεις μας τις εμπορικές, στηριζόμαστε κυρίως στις εμπορικές σχέσεις τύπου εταιρικού, όχι corporate απαραίτητα, αλλά εταιρικές σχέσεις με προσέγγιση ανταγωνισμού. Και αυτό κάνουμε γιατί είναι παρούσα αυτή η μορφή των σχέσεων και στο εσωτερικό του ομίλου και στις σχέσεις με τους εταίρους και στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με το χώρο της γεωργίας και των παραγωγών. Τα προϊόντα λοιπόν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εγγράφονται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για τη διαφοροποίηση, διότι έχουμε πολύ μεγάλα, πολύ πολύ μεγάλα καταστήματα. 8.500 τετραγωνικά μέτρα κατά μέσο όρο έχουν τα σούπερ μάρκετ μας, τα υπερ σούπερ μάρκετ μας και η πεποίθησή μας και η βούλησή μας είναι να αναπτύξουμε ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα καταστήματά μας. Για να μερικά στοιχεία. Σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 30 50% των προμηθευτών και με τη μάρκα τους μπορούν να φτάσουν, με, τις, με τα σήματά τους μπορούν να φτάσουν στο 20% του κύκλου εργασιών μας. Όταν μιλούμε για σήμα λιανεμπορίου, γιατί ξέρετε το 1 τρίτο των, ε, ε, του κύκλου εργασιών μας γίνεται με τη δική μας μάρκα, με το δικό μας σήμα. Το 75% όμως του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Γαλλίας είναι από τις, προέρχεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό και ιδιαίτερο ρόλο μπορούν να δερματίσουν οι μικρομεσές επιχειρήσεις στο φάσμα προσφοράς μας. Για να το εμπλουτίνουμε λοιπόν αυτό το φάσμα προσφοράς προϊόντων, ε, προτείνουμε και ιδιαίτερες υπηρεσίες, όπως πολύ πρόσφατα ένας νέος μηχανισμός που προτείναμε, που προτείνουμε για τη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και σύντομα και την Πορτογαλία, που μας επιτρέπει να δούμε ταχύτατα τους εμπορικούς εταίρους, ε, κατά βάση μόλις μας ε, ε, καταθέσουν το τιμολόγιο τους και φαντάζεστε πόσο πόση σημασία θα έχει αυτό για τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις όταν ε, η ρευστότητα είναι περιορισμένη κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό ως προς την ανταγωνιστικότητα να πτήσουμε τις λεγόμενες φιλιέρ, δηλαδή αλυσίδες επικοινωνίας και προμήθειας προϊόντων με εταιρικέ σχέσεις ισορροπημένες που στόχο έχουν να υποστηρίξουν την τοπική παραγωγή στην εκτινοτροφία, την αλληλεία αλλά και στα οποροκυπευτικά ακολουθούμε αυτή την μέθοδο. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με την προαγωγή μιας προσέγγισης πιο ισότιμης και της ε, ανάγκης που υπάρχει να ξεπεράσουμε τις παραδοσιακές, ε, τους παραδοσιακούς διαχωρισμούς μεταξύ πολύ μεγάλων αγοραστών και πολύ μικρών προμηθευτών. Και γιατί, γιατί πέραν του κύκλου εργασιών και του μεριδίου αγοράς ε, και άλλα κριτήρια επηρεάζουν την αγορά. Υπάρχουν λοιπόν άλλες λύσεις όπως προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση, ανταγωνιστικότητα κτλ. Οι πρακτικές, οι εμπορικές πρακτικές που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μη ε, ισότιμες ή μη ε, Ε, αφήνουν χώρο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ασκήσουν πίεση με το, διαπραγματευτική τους, με διαπραγματευτικό τους ειδικό βάρος και τη δυνατότητα να απαντήσουν πολύ συγκεκριμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών. Και γιατί, διότι και πέραν των εθνικών αγορών, όταν μιλούμε για τα τρόφιμα κυρίως ή τα ποτά, οι αγορές είναι επί το τοπικές. Και βεβαίως, ναι, μπορεί να έχουμε και εισαγωγές και από μακριά προϊόντα, αλλά ε, πάνω απ' όλα έχουμε να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στις ανάγκες των πραγματικά μικρών επιχειρήσεων και έτσι οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δώσουν απάντηση στα συγκεκριμένα συγκεκριμένες ανάγκες είναι αυτές οι οποίες θα ωφεληθούν περισσότερο. Και πολύ σύντομα θα ήθελα να σημειώσω ότι στις εμπορικές μας συναλλαγές προτείνουμε ανάλογα με το μέγεθος ένα σύστημα διαπραγμάτευσης πολύ πιο ελαφρύ για τις μικρές επιχειρήσεις από ό,τι για τις μεγάλες. Στον τρόπο εργασίας μας επίσης έχουμε και συμβάσεις νομικές, πιο απλές, γιατί ξέρουμε ότι η νομική διάσταση είναι πιο δύσκολη βέβαια στο να τη χειριστεί κανείς και έχουν πλεονέκτημα οι μεγάλε επιχείρησει σχέση με τις πιο μικρέ. Επίση, αν χρειαστεί να καταγγείλουμε κάποια σχέση, λαμβάνουμε υπόψη και την ιστορική συνέχεια των σχέσεών μα με κάποιε μικρομεσαίες επιχειρήσει για να επιλέξουμε την ημερομηνία καταγγελίε. Έτσι λοιπόν λαμβάνουμε όλη, μέρημνα για όλα αυτά τα θέματα. Δεύτερη, τρίτη παρατήρηση, η τοποθέτηση του ομίλου σε σχέση με την ρύθμιση των εμπορικών συναλλαγών σε όλη την αλυσίδα. Καταδικάζουμε τις μη θεμητές και μη ισότιμες πρακτικές σε όλη την αλυσίδα, το είπα και την αρχή. Η ρυθμιστική παρέμβαση δεν είναι η κατάλληλη λύση. Η δική μας πρωτοβουλία είναι η σωστή προσέγγιση, πιστεύουμε. Και γιατί. Διότι πολλές χώρες ήδη έχουν σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και επομένω το να εισαχθεί ένα επιπλέον νομοθέτημα δεν αρκεί. Ε, πρέπει όμως να εφαρμοστούν οι νόμοι εκεί όπου υφίστανται. Και τώρα νομίζω αυτό είναι το υπαριθμόν ένα μέλημα. Είτε πρόκειται για εργασία είτε όχι. Εφαρμογή των υφισταμένων νόμων. Επίσης, κάθε ρύθμιση θα πρέπει να δώσει περιθώριο για δημιουργία ε, ε, δέχεται να δώσει περιθώριο για δημιουργία ανε, ανελαστικών σχέσεων, οι οποίε είναι εις βάρος των πάντων. Το που θα πρέπει να κάνουμε θα είναι να δώσουμε, να εξασφαλίσουμε ευέλικτες σχέσεις για να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε, για να μπορεί ο καθένας από τους φορείς και τους δραστηριοποιούμενους στην αγορά να έχει και την σωστή και δίκαιη ανταμοιβή για τη δουλειά του. Επίσης πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν ε, πολιτικές εξουσίες, όποιες είναι αυτές, αποφασίζουν να εισαγάγουν νέους φόρους, διαμεσολάβηση και το καθεξής. Πολύ πρόσφατα στη Γαλλία, το Μάιο συγκεκριμένα, έγινε διαμεσολάβηση για την τιμή του γάλακτος προς όφελος του παραγωγού. Αυτή η διαμεσολάβαση οδήγησε σε αύξηση της ε, τιμής του γάλακτος στο ράφι κατά 5% και αυτή τη στιγμή μειώνονται κατά 11% οι όγκοι κατανάλωσης γάλακτος στη Γαλλία. Γιατί? Διότι υπήρξε άμεση επίδραση στην, αγορά, στην αγοραστική δύναμη του Γάλλου καταναλωτή, ο οποίος περνάει τεράστια κρίση σε πολλές χώρες και ιδίως στη Γαλλία. Αυτά τα συμπεράσματα λοιπόν για να φτάσουμε στην τελική κατάληξη και να σας εξηγήσω στο γιατί ε, υιοθέτησε την, εκούσια, την αυτοδέσμευση και την εκούσια πρωτοβουλία η ομάδα ΟΣΟ, ο οποίο οποίος έχει θεσπίσει κατάρτιση για όλους τους αγοραστές του, δημιουργώντας το 2012 ένα πανεπιστήμιο προσφοράς και ζήτησης, για τους 3.000 ε, αγοραστές ανά τον κόσμο. Ενός πανεπιστημίου λοιπόν όπως το ονομάζουμε, το οποίο έχει ένα μάθημα αγορά ηθική, υπεύθυνη και δεοντολογική για τον Όμιλο Οσό. Αυτό κάνουμε λοιπόν, αγορα... Ε, ορίσαμε έναν διαμεσολαβητή, τον κύριο Μικρομεσαίο, ο οποίος έχει απευθείας επικοινωνία με τον Γενικό Διευθυντή της κάθε χώρας και αποτελεί τον αναπομπό, τον αναμεταδότη των ε, όποιων ζητημάτων ε, πρέπει να υποβληθούν στην προσοχή του. Αυτά για την αγοραστική δύναμη και είμαστε πεπισμένοι σήμερα ότι για να θεσπιστεί αυτό το πλαίσιο εργασίας πολλά ακόμα μένουν να γίνουν, πολλοί χρόνος χρειαστεί. Η κρίση σήμερα μας υποχρώνει να ακολουθήσουμε αυτή την επιλογή. Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που κάνετε. Και υπήρχε και ανταπόκριση. Νομίζω ότι βγαίνουν πολλά μαθήματα από αυτά που λέτε και για τους, αυτούς που διαμορφώνουν την πολιτική. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν πιο ε, χαλαρές σχέσεις... Ε, που να βασίζονται γύρω από τη Σύμβαση ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να τα λάβουν υπόψη αυτά. Θα δώσω το λόγο και στην Κλέρ, η οποία ακούει πάρα πολύ προσεκτικά από το γραφείο του κύριου Μπαρνιέ. Και τώρα ο εκπρόσωπος, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΠΑ Chairman, Ladies um, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ευρωβουλευτές, με μεγάλη χαρά είμαι σήμερα ενώπιόν σας. Μετά τα τελικά συμπεράσματα της ε, Τρίτης το βράδυ για τα κείμενα των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, θα με βλέπετε πολύ συχνά εδώ. Μία από τις βασικές αλλαγές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ είναι ότι εμείς στην ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ ε, εργαζόμαστε για να λάβουμε υπόψη μας ε, τι πρέπει να δώσει αγορά, να κάνει αγορά για τους γεωργούς και τις, τους συνεταιρισμούς. Θέλουμε και αυτός να είναι ένας βιώσιμος οικονομικός τομέας. Θέλουμε να υπάρξουν ε, νέες ευκαιρίες στην χάρη στην εσωτερική αγορά και για τους καταναλωτές επίσης. Η οργάνωσή μας εκπροσωπεί έναν άλλο τομέα που δημιουργεί απασχόληση. Στην Γεωργία έχουμε 25 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 χωρών. Ε, απασχολούμενοι στο λιανεμπόριο επίσης Έχουμε πολλούς, 18 εκατομμύρια συγκεκριμένα ανθρώπους. Επίσης, ε, δραστηριοποιούμαστε στις, ε, στην Ήπεθρο και οι δραστηριότητες μας έχουν τοπικό χαρακτήρα. Υπάρχουν πολύ λίγοι τομεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που, που θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν την γεωργία, ειδικά στις απομονωμένες περιοχές όπου υπάρχει μεγάλο, μεγάλη ανεργία. Το catering και το λιανεμπόριο θα είναι η βασική μας εταίρη για να δώσουμε τα προϊόντα μας στους καταναλωτές. Και επομένως δεν έχουμε καθόλου αυταπάτες για, τις, για τη μελλοντική πραγματικότητα. Θα πρέπει η ευρωπαϊκή διατροφική αλυσίδα να είναι ποιοτική για να δίνει αυτά που θέλει ο κάθε εταίρος της αλυσίδας. Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης και γι' αυτό χαιρετίζω αυτά που είπαν κάποιοι ομιλητές ότι αυτά τα δύο είναι κοινό μας συμφέρον. Όλοι συμφωνούμε επίσης ότι υπάρχουν όντως αφέμητες εμπορικές πρακτικές και το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε σε μια μηδενική ανοχή, αν τα καταφέρουμε να φτάσουμε. Ένα ιστορικό πλαίσιο να θέσω καταρχάς και να πω ότι αναγνωρίζουμε τη δουλειά που έκαναν, Έκαναν διάλογος, πολυμερής διάλογος των ε, ενδιαφερομένων, των stakeholders, όπου είμαστε μέλος και θέλουμε να συμφωνήσουμε σε, ένα, σε μια δέσμη κανόνων για τις ε, πρακτικές, τις εμπορικές σχέσεις. από την αρχή ήταν έντονη η συμμετοχή μας και πιστεύουμε ότι αυτή η δουλειά, αυτό το, αυτή η συζήτηση πρέπει να έχει αποτελέσματα. Συμφωνούμε με αυτή τη δέσμη αρχών. Δεν συμφωνούμε όμως με το καθαρά εθελοντικό πλαίσιο που επιλέχθηκε για να εφαρμόσει αυτές τις αρχές. Ακούστηκε πολλές φορές σήμερα το απόγευμα, πρέπει να, ξεκαθ... εξασφαλίσουμε την εφαρμογή των κανόνων. Στις ε, συζητήσεις της, τελευταίας, της περασμένης χρονιάς και με βάση την εμπειρία των μελών μας, είπαμε ξεκάθαρα ποιες είναι οι ανησυχίες μας σε ό,τι αφορά την ανωνυμία και τις κυρώσεις. Ζητάμε μια νομική γνωμοδότηση που θα λέει ότι χρειαζόταν η νομοθεσία για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες μας σε αυτούς τους δύο τομείς. Οι διατάξεις του εθελοντικού πλαισίου δεν ήταν επαρκείς. Πιστεύω ότι υπάρχει παραπληροφόρηση γενικά σε ό,τι αφορά τη θέση κόπα κοζέκα. Υπόθηκε ότι μόνο νομοθεσία θέλουμε. Μετά την τελευταία μεταρρύθμιση της, ΚΑ, της ΚΑΠ δεν θέλουμε τις βασικές αρχές να τις εμπεριέχουν τα νομικά κείμενα, τα νομοθετικά κείμενα. Δεν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να καλύπτει όλες τις πτυχές της ε, διατροφικής αλυσίδα. Όχι. Αυτή είναι η σκέψη μας. Και μην την ε, διαστρεβλώνετε. Πιστεύουμε ότι όμως ε, και στην αλευθεία του εμπορίου και στις λειτουργούσες, εύρυθμα λειτουργούσες αγορές και στα καλά συμβόλαια, καλές συμβάσεις. Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα πλαίσιο. Ε, υπάρχει σε κάποια κράτη-μέλη, πιστεύουμε στην εσωτερική αγορά, θέλουμε να λειτουργήσει καλά και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρί τη σχετική νομοθεσία. Γιατί δυστυχώ άνθρωποι είμαστε. Και επομένω, θέλουμε ένα μεικτό σύστημα που θα συνδυάσει και νομοθεσία και εθελοντικού κώδικε που θα εφαρμόζονται, τόσο το σύστημα να είναι αξιόπιστο. Και μεγάλη χαρά Ακούσαμε αυτά που παρουσιάστηκαν νωρίτερα από τον κύριο Ντεγιόν και την εκθεσή του, ειδικά για το θέμα της εφαρμογής των κανόνων. Δεν θέλουμε μία άκαμπτη νομοθεσία. Θέλουμε νομοθεσία που θα εξασφαλίσει στους γεωργούς αν προκειμένου και στις, τους συνεταιρισμούς ότι μπορούν να λειτουργήσουν και να είναι προστατευμένοι απέναντι στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και παράλληλα να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί εκπροσωπούμε 38.000 ε, συνεταιρισμού στο γεωργικό τομέα. Οι περισσότερες από, αυτές, από αυτούς τους συνεταιρισμούς είναι μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Ε, οι περισσότερες δε γεωργικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις των γεωργών, είναι μικρές, πραγματικά μικρές επιχειρήσεις. Συνεργαζόμαστε με την κυρία Άλγκρεν για να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι μικρές επιχειρήσεις είναι και αυτές βιώσιμες στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης συνεργάστηκα ε, στα πλαίσια μιας ομάδας για το διοικητικό άχθος. Θα το ξέρετε πολύ. Επίσης ε, θα διαβάσατε την πρόσφατη πράσινη βίβλο. Μόνο με νομοθετικά μέτρα και αποτελεσματική εφαρμογή και προστασία ε, των όσων έχουν παράπονα ε, μπορούν οι αθέμητες πρακτικές να πάψουν να υπάρχουν. Από την εμπειρία που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο προκύπτει ότι οι κώδικες στην διατροφική αλυσίδα άρχισαν να δίνουν αποτελέσματα για τους καταναλωτές και τους λιανεμπορίους αν υπάρχει πραγματική εφαρμογή και έλεγχος. Για να σας πείσουμε και για να κάνω μια ποσοτική αξιολόγηση της οικονομικής επιτύπτωσης των θέμητων εμπορικών πρακτικών στον διατροφικό και γεωργικό τομέα, εμείς ζητήσαμε να γίνει μια ανεξάρτητη μελέτη σε αυτό το θέμα. Και θα σας μιλήσω για τα βασικά πορίσματα αυτής της μελέτης. Πρώτον, όσοι απάντησαν είπαν ξεκάθαρα ότι είναι εκτεθειμένοι σε αυτές τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. 93% των ατόμων που απάντησαν είπαν ότι επηρεάστηκαν τουλάχιστον από μια τέτοια αθέμητη πρακτική. Αυτές οι πρακτικές ε, εμφανίζονται σε όλες τις μορφές εμπορίου και 44% των ατόμων που απάντησαν είπαν ότι εμφανίζονται κυρίως μετά τη σύναψη της σύμβασης, κάτι που προφανώς είναι απαράδεκτο. Επίσης θεωρούν ότι είναι πολύ πιο εκτεθειμένοι σε τέτοιες πρακτικές και από ό,τι ήταν πέντε χρόνια πριν. Σήμερα λοιπόν πιο εκτεθειμένοι από ό,τι πέντε χρόνια πριν. Πάνω από το 50% είπαν επίσης ότι το σημερινό ε, νομικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπίσει αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Επίσης, υπάρχει ε, μία μείωση του κύκλου εργασιών του του κλάδου μας ε, κατέτος 11% ε, με βάση την ε, έρευνα που έγινε. Αυτά που θέσαμε πέρυσι ως ανησυχίες δεν έχουν επιληθεί και νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε σήμερα, αλλά και αργότερα να το συζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα. Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να ξεχάσουμε όλη την καλή δουλειά που έκανε η ομάδα των stakeholders. Εξάλλου δεν πιστεύουμε ότι μόνο οι θελοντικές ε, συμφωνίες ε, είναι αποτελεσματικές. Πρέπει να έχουμε ένα μεικτό σύστημα εθελοντικό και νομοθετικό, ούτως ώστε να δουλεύει το πράγμα καλά. Η ΚΟΠΑ η Ευρωπαϊκή Γεωργή και οι Ευρωπαϊκοί Συνεταιρισμοί είναι ανοιχτή σε διάλογο με όλους τους εταίρους στην ε, διατροφική αλυσίδα. Όπως σας είπα, ο διάλογος είναι ο τρόπος για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Πιστεύουμε ότι η διατροφική αλυσίδα και γενικά το λιανεμπόριο θα δώσει αυτή την ε, προστιθέμενη αξία που θα προσθέσει και θα επαυξήσει το εισόδημα των γεωργών. Του χρόνου είναι το Διεθνές Έτος για τις οικογένειες των γεωργών. όχι, την οικογενειακή, συγγνώμη, γεωργία. Ε, πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια εύρυθμη διατροφική αλυσίδα, συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι οι συμμετέχοντες. Συγχαίρω ξανά τον κύριο Γιόν για την έκθεσή του και ελπίζω ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία ανέφερα θα ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Good. Well, thank you. Uh, Σας ευχαριστώ και τους τρεις. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα το όσα ακούσαμε και πάλι βλέπουμε ότι και πάλι υπάρχουν νέα σχόλια επί της συζήτησης. Ε, μιλήσατε και για το βρετανικό πρότυπο που είναι μάλλον υβριδικό. Λοιπόν, να δώσουμε τώρα τη δυνατότητα στα μέλη να θέσουν ερωτήσεις. Η κυρία Γουλά. <laughs> Πολύ σύντομα, ένα ερώτημα. Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι εξαιρετικά καλή. Όπως είπε και ο τελευταίος ε, ομιλητή είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν και οι γεωργοί σε αυτό το project. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα. Στο λιανικό εμπόριο πολλές φορές αναφέρεται όρους κρίση εγώ θεωρώ ότι δεν μιλάμε αρκετά όμως για την αηφορία σε ό,τι αφορά την ε, χρήση ενέργειας, μεταφορών, πόρων, αλλά και τη βιωσιμότητα σε ό,τι αφορά την, ε, τα απορρίμματα και τη διαχείρισή τους. Ε, είναι και αυτός ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Το ερώτημα μου είναι, εξετάζετε αυτό θέμα στις επιμέρους συμβάσεις σας και ούτω καθεξής. Θέλετε να κάνετε κάτι, γιατί είναι και το οικονομικό σας συμφέρον, αλλά και προς όφελος των ε, καταναλωτών και των πολιτικών να έχουμε μακροπρόθεσμα μία αηφόρο οικονομική ανάπτυξη. Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Uh, Ευχαριστούμε. Ναι, η συμπρόεδρος, Ροξάνα. Ευχαριστώ. Ροξάν Φέλερς ε, ονομάζομαι εργάζομαι για την Food Drink Europe, αλλά εδώ μιλώ με την ιδιότητα της συμπροέδρου μαζί με τον συνάδελφο Ροντρίγκο. Να σα δώσω κάποια πιο ποσοτικά ε, στοιχεία, αλλά να αναφερθώ και στα βασικά συστατικά, αν θέλετε, που οδήγησαν ε, στην επιτυχία της πρωτοβουλίας μας. Να αναφερθώ επιγραμματικά σε κάποια στοιχεία. Διάλογος ο διάλογος ήταν πολύ σημαντικός. Μιλήσαμε πάρα πολύ, αναρρύθμιτες συζητήσεις μέσα σε δυόμιση χρόνια. Θα χρειαστήκαμε χρόνο, είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Μετά, εμπιστοσύνη. Χάρη σε αυτό το διάλογο και το χρόνο αποκτήσαμε εμπιστοσύνη, βασιστήκαμε στην συνένεση και το συμβιβασμό. Φανταστείτε ότι όταν ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, ο καθένας κοιτούσε προς μια άλλη κατεύθυνση τα επιμέρου μέλη της αλυσίδα. Μετά στρέψαμε το βλέμμα ο προ τον άλλον. Και τώρα κοιτάμε, κοιτάμε προς την ίδια κατεύθυνση. Ε, κάναμε πολλά βήματα, καταλήξαμε σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι δεν πρόκειται για πανάκια, όμως πιστεύουμε ότι όσοι συμμετέχουν και βλέπουμε ήδη ότι από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά ήδη έχουμε περισσότερα μέλη. Θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία. Θεωρούμε ότι είναι μία από τις λύσεις που έχουμε στη διάθεσή μας. Και είναι ένας ε, τρόπος ε, να διαχυθεί η προσέγγισή μας ε, στις επιχειρήσεις. Και αυτή η αμφίδρομη προσέγγιση σίγουρα θα μας βοηθήσει στο μέλλον. Αυτά θέλω να πω σήμερα. Ευχαριστώ. Well, thank you very much, and thank you very much for your work on this as well. Yes, now they. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλα ονομάζομαι. Έχω ένα ερώτημα που ε, εμέσως ε, αποτελεί και πρόταση προς την Επιτροπή. Σε μία από τις πρόσφατες συναντήσεις του Governance Group ε, της πρωτοβουλίας τροφικής αλυσίδας, ε, προσκαλέσαμε τον Εθνικό Διαμεσολαβητή της Γαλλίας για τις επιχειρήσεις. Με μια εξαιρετική λοιπόν παρουσίαση μας είπε ότι υπάρχουν, διαχειρίζονται εκατοντάδες επιχειρήσεις, μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων κυρίως, με ένα τεράστιο ποσοστό επιτυχιών μέσα σε τρεις ε, μήνες και μόνο. Το ερώτημα μου είναι μήπως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι η Επιτροπή, η ΙΜΚΟ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνουν ε, την χρήση αυτού του εργαλείου και αλλού. Γιατί ε, έμαθα ότι πρόκειται για ένα μοναδικό παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως... Ε, α, να σας πω επίσης ότι πρόκειται, είναι δωρεάν διαμεσολάβηση. Σίγουρα αυτό θα μα βοηθήσει να επιλύσουμε διαφορέ μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Um, my name is Juan Juan ονομάζομαι. Εργάζομαι για μια ε, ισπανική οργάνωση. Αν δεν σας πειράζει θα μιλήσω ισπανικά, είναι καλύτερα για μένα. Η οργάνωσή μου εκπροσωπεί 4.000 συνεταιρισμού. 96% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στηρίζουμε πλήρως ε, την προσέγγιση της Coca-Cola για έναν ε, πολύ απλό λόγο. Στην Ισπανία ξεκινήσαμε μια παρόμοια πρωτοβουλία, όμως ε, αυτή η πρωτοβουλία πέτυχε ικτρά σε άλλες χώρες, όπως την Πορτογαλία, την Αγγλία και την Πολωνία. Έχουν ξεκινήσει παρόμοιες πρωτοβουλίες και εκεί απέτυχαν παταγωδός. Πολύ απλά γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και οι γεωργοί και οι προμηθευτές, δεν ε, καταδικάζουν ή δεν καταγγέλουν περιπτώσεις ε, αθέμητων πρακτικών γιατί φοβούνται τις επιπτώσεις. Και δεν υπάρχει κάποιος ανεξάρτητος διαμεσολαβητής που να διασφαλίζει την εφαρμογή των αρχών. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν στην Ισπανία δεν θέλουμε να χάσουμε άλλο χρόνο. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό κανονισμό που θα διέπει τις συναλλαγέ μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων. Σε κάποιε χώρε πάνω το 5% ε, των συναλλαγών που αφορούν τα τρόφιμα και ποτά ε, πραγματοποιούνται από αυτού του μεγάλου ομίλου. Όμω, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει πολύ συχνά ε, πλήττονται, δεν μπορούν να προστατευτούν γιατί δεν υπάρχει η απαραίτητη νομοθεσία. Ναι, βεβαίως, να προωθήσουμε τον διάλογο, αλλά Α μην ε, πληγούν και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Σα ευχαριστώ. Πολύ σαφή όλα αυτά. Και αντιλαμβανόμαστε ασφαλώ τα θέματα. Κανείς άλλος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, εάν θέλουμε να επανέλθουμε στον δρόμο της ε, αντιπαράθεσης, θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που πρότεινε ο Ισπανός φίλος και εγώ θα ήθελα να απαντήσω στη δήλωση του κυρίου Πέσσονεν για να πω ότι είναι προσβολή το να λέει κανεί ότι δεν έχει γίνει καμία πρόοδο από το που σηκώθηκα το τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν από 9 μήνε. Έχει συμφωνηθεί ένα πλαίσιο, 450 επιχειρήσει το έχουν προσυπογράψει. Και υπάρχουν όλα τα στοιχεία, άλλωστε τα έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που δείχνουν την υλοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τους μηχανισμούς υλοποίησης και πιστεύουμε, κατά βάση, ότι θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο και με τους διάφορους ε, μηχανισμούς, ε, όποιοι είναι αυτοί, να δίνουμε τις λύσεις. είπε ο συμπροέδρος ότι θα πρέπει να εισαχθεί η κουλτούρα του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης για να αποφεύγουμε τις ε, συγκρούσεις. Η πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει και το ΟΣΟΝ και το Καρφούρ σας τα είπανε, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν αυτά από την μια μέρα στην άλλη αν δεν αλλάξετε στάση συμπεριφορά. Όταν έχετε χιλιάδες αγοραστές και πολλούς περισσότερους εργαζομένους χρειάζεται χρόνος για να γίνει αλλαγή. Η Κόπα Κόζεκ έχει το περιθώριο να επιδείξει ηγετική στάση και θα συνιστούσε να αναλάβει αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Καλά λέει ο πρόεδρος, δεν χρειάζεται να ξέρει αυτή τη συζήτηση. Το Ισάν μας είπε πώς ε, εφαρμόζονται αυτές οι συμφωνίες. Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν διαφορετικούς μηχανισμούς. και θα δούμε αναλόγως πώς θα τους χειριστεί ο καθένας ε, με τις δυνατότητες προσφέροντας στην κάθε χώρα. Σας ακούσουμε όμως την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Συνεργάζομαι τον Επίτροπο Μπαρνιέ στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα. Είπε και η Επιτροπή, ο Επίτροπος μάλλον στην ομιλία του ότι ενθαρρύνουμε μια σειρά από ε, φορείς της αγοράς να ενσωματωθούν σε αυτές τις προσπάθειες, ε, σημειώνοντας φυσικά τις επικρίσεις που ακούγονται, όπως και σήμερα άλλωστε. Αλλά το μέλημά μας είναι να ε, εξασφαλίσουμε εμπιστοσύνη στην αγορά, να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη στην αγορά και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε καινούρια συστήματα για το κάθε τι. Υπάρχουν ε, καλά λειτουργούντα συστήματα στα κράτη-μέλη, μπορούμε να τα συνδυάσουμε με νέα συστήματα. Είπε ο Επίτροπος λοιπόν ότι το ζήτημα δεν είναι η αυτορύθμιση ή η επιβολή κανονιστικών ρυθμίσεων. Υπάρχουν υβριδικά ή μεικτά συστήματα όπως αυτό του γαλλικού παραδείγματος που ακούστηκε νωρίτερα και με την παρουσίαση άλλωστε το είδαμε αποδεικνύει ότι μπορούν να υπάρξουν και να συνυπάρξουν μεικτά συστήματα στην πράξη ωστόσο αυτό σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς ε, θα αξιοποιούν πρώτα τους εκούσιους μηχανισμούς και μόνο αν παραστεί ανάγκη τους ρυθμιστικούς. Βεβαίως και θέλω να ακούσω τι έχουν να πούν οι πρόσωποι εδώ των φορέων για τις ανεξάρτητες αρχές. Βεβαίως και θα κάνουμε εμεί τις προτάσει μας με την αξιολόγηση, η οποία όμως δεν θα κλείνει το βιβλίο αυτής της υπόθεσης, θα αποτελεί μόνο ένα στιγμιότυπο της κατάστασης και θα καταγράφει πόσο αποτελεσματική είναι η... Ε, πόσο αποτελεσματικό είναι το σύστημα και τι ακόμα χρειάζεται να γίνει. Θα ήθελα λοιπόν για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Να πω πόσο σημαντικό το βρήκαν ορισμένοι από τους ομιλητές, αντίστοιχα και εμείς με την περσινή μας ανακοίνωση για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ε, όπου αναφερόμασταν και σε διαφόρους φραγμούς, φορολογικούς και λοιπούς, και που εντωμεταξύ έχουμε ε, ρυθμίσει ε, το βρίσκουμε λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να δούμε όχι μόνο το χώρο των πωλήσεων αλλά και των μεταφορών και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του το έχουμε ρυθμίσει και αυτό. Αλλά πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια ευρύτερη συζήτηση για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στο πρόγραμμα δράσης βλέπουμε ότι, υπάρχει ευρύ, ότι έχει ε, ευρύτερο αντίκτυπο σε όλο τον τομέα του λιανικού εμπορίου. Επίσης αναφέρθηκαν οι τα εμπορικά καταστήματα. Και αν ήταν εδώ ο Επίτροπος Μπαρνιέ θα σας έλεγε ότι είναι προτεραιότητά του το να διατηρήσει την ποικιλία που υπάρχει. Αλλά η οδηγία των υπηρεσιών μας λέει ότι μόνο όταν υπάρχει ε, δοκιμή οικονομικών μόνο στο κοιμή Οικονομικών Αναγκών καταγράφεται, ή καταγράφονται αυτές οι ανάγκες. Βέβαια τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν μια αξιολόγηση και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά η απόφασή τους θα κρυθεί από την αναλογικότητα και την αιτιολογία της. Πρέπει λοιπόν να δούμε και την αναλογικότητα και τα καλά παραδείγματα που μπορεί να υπάρχουν από το ένα κράτος στο άλλο ε, και έτσι θα έχουμε μια πιο σαφή και ξεκάθαρη εικόνα για τι συμβαίνει. Διαπιστώνουμε επίση ότι πολλά πράγματα μένουν να συζητηθούν στο, στην ομάδα υψηλού επίπεδου που έχει δεσμευθεί να θυσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπληρωματικά προ τη δουλειά που γίνεται πέραν τη σημερινή συζήτηση και του χρόνου πάλι με το καλό θα δούμε τι καινούριο θα έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές, όλους τους ελευμένους στη συζήτηση και προχωρώ τώρα στις καταληκτικές παρατηρήσεις καλωσορίζοντας και πάλι την κυρία Γνώρεκα είναι. Με συγχωρείτε, αλλά ακόμα δεν μπόρεσα να μάθω λιθουανικά. Με χαρά σας βλέπω εδώ. Σήμερα η Λιθουανία έχει και την Προεδρία αυτό το εξάμεινο και ξέρουμε ότι πολλά ζητήματα θα τα συστήσουν οι ίδιοι οι Πρωθυπουργοί ή καλύτερα Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί του Ευρωπαϊκού Συμβούλου για να μην πιο σαφής. Γι' αυτό αν έχετε την καλοσύνη να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάρμπορ. Αγαπητή κυρία Κοράτσα Βίλτ, αγαπητή βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εδώ παριστάμενοι εκπρόσωποι του κλάδου, με μεγάλη χαρά είμαι εδώ σε αυτή την εκδήλωση. Είναι πολύ σημαντικό για την Λιθουανική Προεδρία του Συμβουλίου να ε, το ότι έχει την ευκαιρία να παρήσετε σε αυτήν την πρώτη συζήτηση του Ρογγυλής Τραπέζι για το ελληνικό εμπόριο και να συνεχί, να βλέπει τη συνέχιση του έργου που ξεκίνησε με το ψήφισμα του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5 Ιουλίου του 2011 και αν μου επιτρέπετε αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα τώρα, μια και προσφέρει αυτή την ε, υπηρεσία το Κοινοβούλιο πολύ ευγενικά, να μιλήσω στη μετρική μου γλώσσα τη λιθουανική. Ε, Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου η Ευρώπη αγωνίζεται να ξεφύγει από την κρίση όπου οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και λοιποί παραγόντες αναζητούν τρόπους για ανόρθωση της οικονομικής ανάπτυξης και την σταθερότητα. Ο χώρος του λιανικού εμπορίου προσφέρει πάνω από 15% όλων των, των συνόλων των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια της κρίσης όμως βρέθηκε σε μια κατάσταση πάρα πολύ ευάλωτη και επλήγει βαρύτατα από την κρίση και στη Λιθουανία, ο χώρος του λιανικού εμπορίου. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είχαμε σημαντική πτώση του κύκλου εργασιών. Ο κύκλος εργασιών του 2010 είχε μείωση, παρουσίαζε μείωση σχέση με αυτόν του 2008 κατά 28%. Αυτό σημαίνει σημαντική συρρήκνωση των οικονομική δραστηριότητα και των θέσεων εργασία. Και βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι και σε άλλα κράτη-μέλη εμφανίστηκαν αντίστοιχα προβλήματα. Γι' αυτό και θα ήθελα να συγχαρώ το Κοινοβούλιο και να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της Επιτροπής και την κυρία Κοράτσα Μπίλτ ε, για την πρωτοβουλία αυτή. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντε ο οποίο αναλαμβάνει τη συνέχιση του έργου που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια και τη συζήτηση αυτού του ζητήματος. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σε συνεχή επικοινωνία βέβαια με τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς ε, ε, δίνουν μια βάση συζητήσεως πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική δεν ήταν τυχαίο το γεγονό πώ ανέφερα ότι το κοινό μα έργο, κοινό έργο όλων των θεσμικών οργάνων, είναι ένα έργο με πολύ μεγάλη σημασία. Στον τομέα του λιανικού εμπορίου φυσικά. Η Προεδρία της Λιθουανίας θα αναλάβει την πρωτοβουλία και θα τοποθετήσει την Ευρωπαϊκή Ενία Αγορά στο επίκεντρο του θεματολογίου για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων Σήμερα έγινε συζήτηση πολιτικής στο Συμβουλίο Ταγωνιστικότητας για την, για την ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Απευθύναμε ερωτήσει ε, στον Υπουργό για το τι μέτρα μπορούν ε, να αναλυφθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσανάλογα ε, ανελαστικοί περιορισμοί και αυτά τα συμπεράσματα από τη συζήτηση θα συμπεριληφθούν στο ε, χρονοδιάγραμμα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας του Δεκεμβρίου. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξέρουμε καλά ότι είναι το 95% των επιχειρήσεων του τομέα της Λιανικής και μόνο 8% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδίονται σε διασυνοριακό εμπόριο, ηλεκτρονικό εμπόριο. Γι' αυτό χρειάζεται όμως η εσωτερική αγορά. Δεν χρειάζεται να κοιτάμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, σε αντιπαράθεση με τις μεγάλες. Πρέπει απλώς να τους αφήσουμε ένα περιθώριο και να τις ενθαρρύνουμε να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους πέραν των συνόρων. Όπως ακριβώς πράττουν και στην ε, χώρα τους έτσι, νομίζω μπορούμε να αναφερθούμε στην ε, καλύτερη εφαρμογή των κανόνων για την ε, αγορά, για τη λιανική αγορά, την εφαρμογή των, των κανόνων της αμοιβέ αναγνώρισης στα κράτη-μέλη και να πούμε ότι ο τομέας του λιανικού εμπορίου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Θα πρέπει όμως να δούμε και την διοικητική πλευρά, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε δηλαδή τις επιχειρήσεις. Αυτό θα καταγραφεί οπωσδήποτε και πιο λεπτομερώς στα συμπέρασμα του Συμβουλίου. Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ομάδα εργασία υψηλού επίπεδου για την ενίσχυση τη αγωνιστικότητα, τι οποίε οι συστάσει θα συμβάλλουν, φαντάζομαι, πολύ στην ενίσχυση τη αγορά ε, λιανικού εμπορίου. Επίσης το έργο της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ και το πρόγραμμα, λεπτομέρειες πρόγραμμα δράσης του κυρίου Ιόγκ θα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις αισθήσεις μας τον Δεκέμβριο. Η λειτουργία της νέας αγοράς βαίνει παραλλήλως με μια ε, καθαρή διαφανή και ισότιμη εταιρική σχέση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και μεγάλη χαρά σήμερα ακούω ότι είναι 450 επιχειρήσεις έχουν προσπογράψει την εκούσια δέσμευση για τον τομέα της λιανικής. Αυτό νομίζω αποδεικνύει πόσο αναγνωρίζουν ότι είναι κατεπίγουσα η ανάγκη να αναλάβουν δράση. Πρέπει λοιπόν να τις ενισχύσουμε, πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε όθηση στις προσπάθειες αυτές και να ενθαρρύνουμε οποιοδήποτε θέλει να συμμετάσχει σε αυτή την εκούσια δέσμευση. Ελπίζουμε ότι έτσι θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την εκδήλωση, η οποία ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα και πηγή αισιοδοξίας Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ευχαριστώ που συνδέεται το έργο της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ με το πακέτο για το λιανεμπόριο. Υπάρχουν και διάφορα άλλα σημαντικά θέματα που ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε, ειδικά για την εποπτεία της αγοράς και, το... και την εποπτεία των καταναλωτικών προϊόντων. Ένα από τα θέματα του REACH είπε κάποιος ομιλητής. Κάτι που μου θύμισε ο εκπρόσωπος Κοπακοζέκα. Δέωσα τη δυνατότητα στους ε, τελευταίους ομιλητές, ε, τους τελευταίους ε, ομιλητές του δεύτερου πάνελ δηλαδή, να σχολιάσουν κάποια από τα πράγματα που άκουσαν. Και εν συνεχεία η κυρία Κοράτσα Μπίλτ θα κάνει τα τελευταία σχόλια. Short interventions, από τους τρεις ομιλητές, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέω ο πρώτος από τους τρεις ομιλητές. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω για το θέμα της εφαρμογής. Γιατί είναι το θέμα. Τα διαφορετικά κρατημέλη βρίσκουν διαφορετικές λύσεις στο θέμα της εφαρμογής. Κάνα πρόβλημα. Αλλά από αυτά που είδα στο governance group και, και τις συζητήσεις που κάναμε, δεν υπάρχει εφαρμογή. Η εφαρμογή στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όταν πρόκειται για εφαρμογή της νομοθεσίας, δεν, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι συμβατή με τις εθελοντικές πρωτοβουλίες. Από τις διαπραγματεύσεις που είχαμε, προκύπτει ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιληθούν οι διαφορές είναι το να αρκεστούμε και να αφήσουμε το πράγμα στο εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό θέλω να ενθαρρύνω τη δημιουργία εθνικών, εθνικής πλατφόρμας και να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσει εκείνες τις υποθέσεις όπου υπάρχει διασυνοριακή διάσταση να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν η εθνική λύση δεν μπορεί να βρεθεί. Επομένως, δεν καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Ισπανός συνάδελφος όταν λέει ότι στην Ισπανία βρήκαμε τη, λύση, στο Ηνωμένο Βασίλειο βρήκαμε τη λύση. Οκ, αλλά τότε γιατί θέλετε να βάλετε και άλλο ένα στρώμα ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τι σκοπό εξυπηρετεί η ευρωπαϊκή λύση, εν πάση περιπτώσει. Merci, <coughs> Ο δεύτερος ομιλητής. Να προσθέσω αυτά που είπε ο προλαλής σας, ότι οι εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις διέπονται από την κουλτούρα, τις αντιλήψεις μας, τις ιδέες μας και μέσα από την πρωτοβουλία που ξεκίνησε τα πράγματα φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη, ότι είναι ρευστά. Και μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται χρόνος για να γίνουν πρακτικές οι διάφορες λύσεις και να τις εφαρμόσουν διάφοροι ενδιαφερόμενοι. Ορισμένες πρακτικές, ορισμένες ε, λύσεις έχουν γίνει πρακτική, αλλά είναι θέμα εμπιστοσύνης και χρειάζεται χρόνος μέχρι να οριμάσουν τα πράγματα. Νομίζω ότι μέσα από το Πανεπιστήμιο ΣΟΝ θα μπορούσατε να περάσετε κάποιες από τις ιδέες σας. Είναι μια νέα, μια φρέσκια ματιά αυτή. Να συμπληρώσω αυτά που είπε ο Χριστιαν. Δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα με τις δηλώσεις μας. Εγώ είμαι Γενικό Γραμματέα Κοβακοζέκα 7 χρόνια. Και από την εμπειρία που έχω, σας δηλώνω ότι Πραγματικά φαίνεται ότι αλλάζουν τα πνεύματα μέσα αυτά τα τελευταία 7 χρόνια. Τον Ιούλιο του 2012 συζητήσαμε αυτά τα πράγματα και υποστήριξαμε την κοινή πρωτοβουλία. Και εγώ είπα ότι πρέπει να εγκρίνουμε αυτή την πρωτοβουλία και να προχωρήσουμε, αλλά τελικά δεν εγκρίθηκε. Δεν εγκρίθηκε από την Κοπακοζέκα, από το Προεδρείο της Κοπακοζέκα. Απέτυχα ως Γενικός Γραμματέας. Είπα να δώσουμε λίγο χρόνο, λίγο περιθώριο. Ε, άλλους 6 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο. Και όπως είπε και η Ροξάν, ναι, δώσαμε αυτό το χρόνο. Αλλά στη συνάντηση του Προεδρείου, το Δεκέμβριο, είδα ο κόσμος να έχει κάνει στροφή 180 μοίρες, σχεδόν όλοι άλλαξαν γνώμη. Δηλαδή, χάρη σε αυτού τους 6 μήνε χρονικού περιθωρίου, άλλαξαν τα συμπεράσματα του Ιουνίου, Ιουνίου όχι του 2012. Δεν είχε εγκριθεί αυτό το θέμα. Υπήρχαν δύο θέματα. Ανωνυμία και κυρώσει. Και μου είπαν, κοίταξε κύριε Γενική Γραμματέα, αυτά είναι δύο τομείς που δεν μπορούν να περάσουν. Παρ' όλα αυτά, εμεί ενδιαφερόμαστε αυτό το σύστημα να δουλέψει. Όχι με άκαντο τρόπο, όμως. Αλλά, Κρίστιαν, πρέπει να ξέρεις ότι η εναλλακτική που μας λες δεν είναι επιτάπητος. Θέλουμε όχι κάτι άκαμπτο, αλλά θέλουμε μια διατροφική αλυσίδα στην Ευρώπη, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι λειτουργούν μέσα σε ένα ρευστό, ας πούμε, πλαίσιο. Το πλαίσιο μας στο οποίο κινούμαστε δεν είναι αποτελεσματικό. Γι' αυτό και είμαστε εδώ σήμερα. Αισθάνθηκα πραγματικά ότι έπρεπε να μιλήσω με εσά, κύριε Πρόεδρε, με τους συναδέλφους. Δεν υπάρχει καμία εχθρότητα. Απλώς ε, αυτό το σύστημα δεν φέρνει, καρπούς, δεν φέρνει τους καρπούς που θέλαμε. Πρόεδρος. Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία και γι' αυτό χαιρόμαστε που ήρθατε εδώ. Είναι μια νέα εμπειρία για μας γιατί δεν είχαμε ασχοληθεί μέχρι τώρα με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ τους Ερμηνείς που μας δίνουν λίγο παραπάνω χρόνο. Να δώσουμε το λόγο ε, στην Αναμαρία. Ευχαριστώ. Ναι, εμένα με κατατοπίζει ιδιαίτερα αυτή η συζήτηση, γιατί ακριβώς αυτό θέλουμε, μια ζωντανή συζήτηση ουσίας ε, με τους πραγματικούς ενδιαφερόμενους ε, και τις εμπειρίες τους. Πήρα τόσες πολλές σημειώσεις που δεν έχω πλέον που να τις βάλω. ακούσαμε με προσοχή και Βεβαίω και θα δοθεί συνέχεια. Εντάξει, όλοι θέλουμε να γυρίσουμε τώρα σπίτια μα, αλλά δώστε μου δύο λεπτά για το ζήτημα αυτό της ε, ισότητα της δικαιοσύνης. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θέλουμε να βρούμε λύσεις που θα φέρουν αποτελέσματα. Με πραγματική δέσμευση. Αυτό που θέλουμε και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, είναι ότι είναι μοναδικό επίτευγμα από μόνο του αυτή η πρωτοβουλία. Ότι βρισκόμαστε εδώ με τους δύο ε, από, τις μεγαλύτερου από τους μεγαλύτερους ομίλους σούπερ μάρκετ της Ευρώπης. Ε, Ροντρίγκο, Ροξάνα, άνθρωποι που ηγούνται των διαπραγματεύσεων και τόσοι άλλοι φορείς και συζητούμε ανοιχτά σε δημόσιο διάλογο, σε σε ένα ευρωπαϊκό όργανο και ο, ο Επίτροπος Μπαρνιέ είπε ότι τα όργανα είναι στη διάθεσή σας, στην υπηρεσία σας και αυτό είναι τμήμα της λύσης. Σας καλώ λοιπόν ε, να συνεχίσετε τις διαπραγματεύσεις. Κατανοούμε ότι το θέμα της ανωνυμίας και των κυρώσεων είναι εξαιρετικά σημαντικά για, τη, τα μέλη σας. Δηλαδή μια μικρή επιχείρηση φοβάται να, να χάσει έναν πελάτη. Αν χάσει ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να μην τα βγάζει πέρα πλέον. Και πρέπει να σταματήσουμε βεβαίω να μιλάμε για, μικρά, για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, να μην ε, δαιμονοποιούμε τις μεγάλες επιχειρήσεις και προστατεύουμε τις μικρές. Ε, πρέπει να προχωρήσουμε από αυτή την προσέγγιση. Κάποιοι φοβούνται λοιπόν να χάσουν ε, Επιχειρηματικού εταίρους, αλλά από εκεί και πέρα χαίρομαι που βλέπω ότι υπάρχει πρόοδος, όχι μόνο στις Βρυξέλλες, αλλά και στην πραγματικότητα, στα κράτη-μέλη. ξεκινάμε από τις Βρυξέλλες, αλλά πλέον κινούμαστε και φεύγουμε και πάμε και προς ε, τις περιφέρειες, ε, τα κράτη-μέλη, τους καταναλωτές. Και Μία από τις ειδήμονες σε αυτό το τομέα δεν είναι εδώ απόψε γιατί δίνει διάλεξη σε, έναν, ε, σε μια οργάνωση αγοραστών ε, σούπερ μάρκετ. Αυτό πριν από δύο χρόνια δεν θα συνέβαινε. Θα ακούγαμε CEOs να έρχονται, διευθύνονται συμβούλους να έρχονται να μας λένε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό θα βλέπαμε. Τώρα όμως ακούστηκε σήμερα ότι υπάρχει πρόβλημα, κάτι πρέπει να γίνει και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Εσάς βεβαίως δεν σας φτάνει. Ακούσαμε όλες αυτές τις απόψεις. Αλλά θεωρώ ότι η απλή μεταφορά ενός συστήματος που μόλις ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία με αυτή τη δυνατότητα μεσολάβησης δεν νομίζω ότι είναι αυτομάτως και μια λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βρούμε ε, κάτι το ενδιάμεσο, δηλαδή εφαρμογή της νομοθεσίας αλλά και εξέταση της πραγματικότητας στα κράτη-μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με εσά βεβαίως για να δώσουμε μια δυνατότητα στην πλατφόρμα με παρακολούθηση, αξιολόγηση, διακυβέρνηση, δομή βεβαίως ε, που καλύπτεται από αυτή την οργάνωση ομπρέλας και μπορούμε να επανέλθουμε εδώ σε ένα χρόνο ή στα άλλα δύο φόρουμ που έχουμε στη διάθεσή μας και εσείς που έχετε τη διάθεσή σας για να ανταλλάξετε απόψεις, να πείτε ότι εκεί τα πήγαμε καλά, εκεί όχι, κάτι έγινε, αλλά πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα για την ανωνυμία και τις κυρώσεις. Έτσι μπορούμε να αποδείξουμε τη δέσμευσή μας. Και η κυρία Υπουργό ε, βρέθηκε και έμεινε μαζί μας όλο το απόγευμα και αυτό είναι δείγμα δέσμευσης και από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ότι θέλουμε να δώσουμε αυτή την ανεξάρτητη δυνατότητα σε εσά για να δούμε αν θα λειτουργήσει ή όχι. Ροντρίγκο, θέλεις χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος. Η πολιτική πίεση είναι μεγάλη. Πολιτική πίεση για να αναλάβουμε δράση. Πρέπει να βρεθεί μια εμπειρία, γιατί εσύ θέλεις χρόνο, από την άλλη δεν υπάρχει χρόνος. Απαιτείται χρόνος για να αλλάξουμε νοτροπίες, αλλά επιχειρήσεις δεν έχουν χρόνο, χρονοκοπούν. Και θα πρέπει να υπάρχει μια αλληλοκατανόηση στο πλαίσιο ενός διαλόγου. Ελπίζουμε να συνεχιστεί, εμείς εκεί θα είμαστε και θα παρακολουθούμε. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, δεν έχω χρόνο. Απλώς εν συντομία να απαντήσω σε μερικά ακόμα σημεία. Στη συνάδελφα Ρούλερ για το ζήτημα της αηφορίας. Δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε πάνελ για την ε, βιωσιμότητα, όμως ε, είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Ε, βεβαίως ξέρετε πόσο με απασχολεί το θέμα της ε, απόρριψης τροφίμων. Έχουμε ακόμα και πλατφόρμες όπου με θελοντικές πρωτοβουλίες ε, των εμπορευομένων της ε, αλυσίδας εφοδιασμού και εκεί έχουμε πολλά αποτελέσματα στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα και στην μείωση των εκπομπών διευθυντήτων του άνθρακα. Και άλλες πρωτοβουλίες για την μείωση των απορριμμάτων. Ε, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου δύο ακόμα σημεία. Το θέμα της πρόσβασης ε, για τους καταναλωτές που ζουν σε πόλεις, πρόσβαση λοιπόν σε ζωντανά κέντρα πόλεων, αλλά και στις απομακρυσμένες περιοχές, είναι ζητήματα που μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως. Και εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερο τρόπο να προστατεύσουμε του μικρού είναι να του δώσουμε τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν. Μέσω τη ανταγωνιστικότητα, όχι μέσω του προστατευτισμού. Πρέπει να ανοίξουμε τι αγορέ. Περισσότερο ανταγωνισμό λοιπόν, όχι περισσότερη προστασία. Έτσι σώζουμε του μικρού και εν μέσω κρίση Είμαι εισηγήτρια και για την ε, έκθεση της, ε, για την οδηγία υπηρεσιών και λέμε ξεκάθαρα ότι είμαστε κατά αυτών των οικονομικών συμφερόντων, όχι γιατί δεν είμαστε υπέρ της επικουρικότητας, πρέπει να υπάρχει ε, αυτή η χωροταξία. Όμως αυτά τα, τα τεστ των οικονομικών ε, αναγκαιοτήτων και αναγκών έχουν ε, χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για να κλείσουν οι αγορές σε επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών. Χρησιμοποιείται λοιπόν για σκοπούς διάκρισης, όχι για την προώθηση της αηφορίας προστασίας του περιβάλλοντος σε πολλές περιπτώσεις. Γι' αυτό και ζητούμε από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και την οδηγία υπηρεσιών για την πρόσβαση στην αγορά με ισότιμους όρους συνταγωνισμού και σε επιχειρήσεις από άλλα, από άλλα κράτη-μέλη. Κύριε Πρόεδρε, προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μου με όλους. Νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος ε, για την Επιτροπή μας να ε, συνεργαστεί και με τους εμπορευομένους της ε, εσωτερικής αγοράς. Σας ευχαριστώ όλους θερμά που βρεθήκατε εδώ σήμερα και όσους συμμετείχαν στη συζήτηση στο Twitter και σε όσους ακούσαν από το σπίτι. Ευχαριστώ πολύ. Well, um, I'd like to, uh, thank all of you. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας και όσους μας παρακολουθούν από το σπίτι. Συμφωνείτε μαζί μου ότι και η συζήτηση στο Twitter σίγουρα προσέθεσε στο ενδιαφέρον της συζήτησης. Χαιρόμαστε που βλέπουμε τέτοιο ενδιαφέρον. Είναι ένα πείραμα που θα συνεχίσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα Twitter εντό εισαγωγικών, δεν ξέρω μπορείτε να αποκολέσω έτσι. Αυτοί μας βοήθησαν όμως, ιδιαίτερα τη Ρίκα. Σας ευχαριστώ και για την πρόταση. Ήταν μια νέα ρεξικέλευθη πρωτοβουλία που πήραμε με την Άννα Μαρία να κάνουμε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα και να επικεντρωθούμε στην πτυχή της εσωτερικής αγοράς και τους καταναλωτές. Την επόμενη φορά καλό θα τα αναφέρουμε περισσότερους καταναλωτές. Αυτή τη φορά έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα να θίξουμε. Βεβαίως μας απασχολεί και η προσέγγιση των καταναλωτών και τι θέλουν εκείνοι σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, την ανταπόκρισή τους σε προσφορές, ε, τις αγοραστικές τους τάσεις ε, και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στους συναδέλφους ε, εδώ που μας παρουσίασαν πραγματικά πρωτότυπο έργο που μας εμπνέει να συνεχίσουμε. Ελπίζω και εσείς να εξετάσετε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την ενιαία ψηφιακή αγορά που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία ε, τον Ιούνιο και, υποβλήθηκε και θα υποβληθεί στον Οικονομική Σύνοδο Κορυφής του επόμενου μήνα όπου θα τεθούν στην εμείς διάταξη τα ζητήματα της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και του καθεξής. Κλείνοντας, μείνετε σε επαφή μαζί μας. Υπάρχουν και αντίτυπα του ενημερωτικού μας δελτίου, αν δεν το έχετε λάβει. Αν δεν είστε στο κατάλογο email μας, βεβαίως μπορείτε να εγγραφείτε για να σας στέλνουμε τακτικά mail. Και θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για να διατηρήσουμε και να πραγματοποιήσουμε την ολοκλήρωση της ενέργειας αγοράς. Και για τους παραγωγούς βεβαίως είναι σημαντικό όλο αυτό. γιατί ε, σήμερα παρευρίσκεται εδώ και μια πολύ σημαντική ομάδα του γεωργικού κλάδου. Της Γεωργικής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους ε, διερμηνείς που μείνατε και λίγο παραπάνω. Καλό απόγευμα.